Ε, Καλημέρα σας, με συγχωρείτε που θα μιλήσω Ιταλικά, για μένα είναι πιο εύκολο. Σας υπενθυμίζω ότι... Ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται με το διαδίκτυο. Περνάμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη, η οποία σας διανεμήθηκε στις 8 Ιουλίου και εάν συμφωνείτε, θεωρώ ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Και υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις. Και να σας πω επίσης ότι είναι η πρώτη φορά που εκτελώ χρέη προέδρου και καταλαβαίνω θα κάνω πάρα πολλά λάθη και αν βέβαια μπορείτε συγχωρήστε με παρακαλώ. Πάμε στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Οι σοσιαλδημοκράτες ενημέρωσαν τη γραμματεία για τον ορισμό ε, της κυρίας Μετσέντες Μπρέσο η οποία θα γνωμοδοτήσει για την έκθεση Επιτροπής Κόντε σχετικά με την έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μάχη κατά της απάτης. Είναι μια γνωμοδότηση που διανεμήθηκε από την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών στην τελευταία συνεδρίασή μας. Εάν λοιπόν θεωρείτε ή συμφωνείτε όλοι, εγκρίνεται αυτός ο ορισμός ε, με επίσης ε, την δική μας επιβράβευση. Πάμε στο τρίτο σημείο. Εκεί θέλω να σας πω ότι υπάρχουν οι συστάσεις των ε, συντονιστών οι οποίοι συνεδρίασαν στις 6 ε, Ιουλίου αυτού του έτους το 2015 στο Στρασβούργο. Οι συντονιστές λοιπόν θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν για την έκθεση την οποία ε, θα προετοιμάσει η Επιτροπή Αναφορών σε σχέση με τις ενέργειες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2014 και οι ίδιοι συγητές ενέκριναν την νέα ημερομηνία που προτείνεται που είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015 από τις 1.30 ε, μέχρι τις 3.30 ε, το μεσημέρι. Εκεί να γίνει μια συνάντηση ε, με μια αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης και αυτή η συνάντηση θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες. Και επίσης επιβεβαίωσαν ότι η Διευκοινοβουλευτική συνεδρίαση της ΑΦΚΟ που η ΑΦΚΟ θα οργανώσει με τις ε, αντίστοιχες επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτή η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίας Επιτροπής ΑΦΚΟ και αυτό 5η ε, 19 Νοεμβρίου του 2015. Αυτή η συνεδρίαση θα γίνει από κοινού με το εργαστήριο το οποίο οργανώνει ε, η υπηρεσία για τα αστικά δικαιώματα συνταγματικές υποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης ΥΠΟΛ. E Εκεί θα εξεταστεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ε, στις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, η αποστολή της ΑΦΚΟ στην Ουάσιγκτον εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων που έλαβε χώρα τον Ιούλιο και αυτή θα γίνει κατά τη διάρκεια της 45ης ε, εβδομάδας. Εβδομάδα ε, Τυρκουάζ είναι η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Επίσης ε, η δική μας Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τις ε, συστάσεις ε, που σας ανέφερα και τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι κλείσαμε και με αυτό το θέμα. Και τώρα λοιπόν περνάμε στην ουσία, στο διατάφτα, Το θέμα μας είναι η βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιώντας το δυναμικό της συνθήκης της Λισαβόνας. Οι συγητές, ως γνωρίζετε, είναι η κυρία Μετσέντες Μπρέσο και ο κύριος Έλμαρ Μπρόκ. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Ποια είναι η άποψή μου επί του θέματος. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα μόνιμο αίτημα. Και υπάρχει κάτι που θέλω να πω σε εσά, το λέω βέβαια και στον εαυτό μου. Εγκρίθησαν τρεις εκθέσεις πρωτοβουλίες σχετικά ε, για τις δυνατότητες που παρέχει η συνθήκη και οι δυνατότητε τη και νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ σημαντική νύχτα για την ιστορία της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Αναφέρομαι στην τελευταία Κυριακή που αφορούν ε, στις προποθέσεις υπό τις οποίες θα παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Κατά την άποψή μου αυτή ήταν μια καταστροφική νύχτα και αυτό κάτω από πολλά πρίσματα και απόψεις. Όχι μόνο για την Ελλάδα η οποία οθήθηκε να δεχθεί μια λιτότητα που ο λαός όμως είχε απορρίψει πλειοψηφικά αλλά ήταν και μία μαύρη νύχτα για τη δική μας την Ένωση. Αυτό λοιπόν που σας καλώ είναι να πείτε με απόλυτη ειλικρίνεια κατά πόσον είναι σωστό να διατηρηθεί αυτή η μερίσια διάταξη με τις δύο εκθέσεις να μην έχει γίνει τίποτα. Ίσως θα ήταν πιο σκόπιμο να μιλήσουμε για τις δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη και να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Να μιλήσουμε Έχοντα κατά νου ότι υπήρξε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο πολλοί το ερμήνευσαν όχι μόνο ως αποφάσεις που με τη μορφή ταπείνωσης ενός ολόκληρου λαού αλλά και κάτω από το πρίσμα του κατά πόσον έχουμε μια ενωμένη και αλληλέγγυα Ευρωπαϊκή Ένωση όπως πολλοί το επιθυμούμε. Πλέον είναι μια Ευρώπη η οποία διατρέχει κίνδυνο να αποσυνδετεί μια ευρωπαϊκή, μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία δείχνει ότι είναι αδιάφορη προς όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται. Η δική μας λοιπόν η Ένωση είναι σαν να είναι ένα φόρουμ ανθρώπων που ομιλούν χωρίς να γίνεται επί της ουσίας κάτι το συγκεκριμένο. Εκείνο λοιπόν το οποίο σας καλώ να πράξετε και εδώ απευθύνομαι κυρίως στους εισηγητές είναι πλέον να συλλογιστούν. Διάλειμμα και περισυλλογή. Καλό λοιπόν όλους σας ε, να εκφράσετε τις απόψεις σας ε, για την ένωση την οποία επιθυμούμε. Μία ένωση η οποία θα είναι διαφορετική από αυτή που έχουμε ακόμα και αν δεν τροποποιηθούν οι συνθήκες και αυτό πρέπει να το κάνουμε αν δεν επιθυμούμε η εικόνα που παρουσιάζει η Ευρώπη προς τους πολίτες να επιδεινωθεί περαιτέρω. Θέλω λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι πέρυσι το Μάρτι είχαμε μία ακρόαση για το θεσμικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από αυτά που αναγράφονται στις συνθήκες. Η δική μας λοιπόν επιτροπή τοποθετήθηκε όσον αφορά την διακυβέρνηση και το θεσμικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια γνωμοδότηση της 19ης ε, Μαΐου, αυτή συντάχθηκε από την ΟΚΕ και από την Επιτροπή των Περιφερειών και σήμερα έχουμε τη χαρά να μπορούμε να δεχθούμε στους κόλπους μας ε, τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, των Περιφερειών, τον κύριο Μάρκουλα, ελπίζω και να πρόφερα και σωστά το όνομά σας, ο οποίος ε, θα μας παρουσιάσει το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών στις 8 Ιουλίου. Αυτό λοιπόν το ψήφισμα δόθηκε σε όλα τα μέλη την ε, Παρασκευή. Ε, Δόκτωρ Μάρκουλα θα σας δώσω το λόγο έτσι ώστε να μπορέσετε και εσείς να μιλήσετε και να ξεκινήσει η δική μας συζήτηση με τη δική σας την εισαγωγή. Ευχαριστώ κυρία Σπινέλη, κυρία Μπρέσκο, κυρία Χέλμαρ Μπρόκ, αγαπητοί ευρωβουλευτές. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι διαβουλεύεστε την Επιτροπή των Περιφερειών για το θέμα της συνθήκης Λισαβόνας και το επέκεινα. Ε, μιλήσαμε για το πώς θα προσαρμοστεί το ψήφισμα Έχετε μπροστά σας την, την πράσινη μπροσούρα όπου τονίζει τις απόψεις του εισηγητή και των βασικών εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων μας. Το ψήφισμα καλύπτει και την έκθεση Μπρέσκο και την έκθεση και την έκθεση του Φερχόφστα που θα προσαρμοστεί μετά. Σας ευχαριστώ για το, την επαφή που είχαμε με τους εισηγητές στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Όλοι συνεισέφεραν. Μοιράσαμε αυτό το φυλάδιο με τα βασικά στοιχεία που αναφέρετε εσείς ε, και τα μέλη μας. Και με μεγάλη χαρά μπορώ να σας μιλήσω για κάποια από τα βασικά θέματα που πιστεύουμε και θα διαιρέσω την παρέμβασή μου σε δύο μέρη. Καταρχάς, τι βήματα μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια των ισχυουσών συνθήκων και δεύτερον τι προτάσει που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε όταν και εφόσον γίνει η μεταρρύθμιση των συνθήκων. Οι βελτιώσει στην ισχύουσα συνθήκη τη Λισαβόνα. Ξεκινάμε με το μοναδικό ρόλο τη συνθήκη τη ε, Επιτροπή των Περιφερειών ω ε, συμβουλευτικό σώμα που εκπροσωπεί τι ε, τοπικέ και τι περιφερειακέ αρχέ. Ο ρόλο μα έχει αναπτυχθεί με κάθε νέα συνθήκη, αλλά ο ρόλο μα στην ε, νομοθετική διαδικασία θα μπορούσε να αναγνωριστεί πιο επίσημα. Η λόγη είναι απλή. Έχουμε μια διπλή νομιμότητα. Καταρχά, μια δημοκρατική μέσω των εκλεγμένων ε, μελών μα από τι πόλει μα και μια νομική που εκπροσωπούμε, τα μέλη μας εκπροσωπούν τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ. Έχουμε νομικές ευθύνες για να εφαρμόσουμε δηλαδή τη νέα νομοθεσία. Και αυτές οι νομικές ε, αποκλειστικές μερικές φορές είναι αποκλειστικές. Μερικές φορές βεβαίως είναι επιμερισμένες με τις εθνικές κυβερνήσεις. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο υπό τις ισχύουσες συνθήκες να καταστήσουμε την ε, θεσμική μας νομιμότητα πιο συμβατή με τη λειτουργία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε το ρόλο των, της των Περιφερειών ούτω ώστε να μπορούμε άμεσα να αξιοποιούμε τη γνώση και την εμπειρία των τοπικών ερετών αρχόντων. Να σας κάνω τις εξής προτάσεις. Καταρχάς, στην αρχική φάση σύνταξης της νομοθεσίας. Εκεί πρέπει να γίνει προσπάθεια. Αυτό έχει συζητηθεί πολλές φορές με τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και αυτό συμπεριλαμβάνει την, μια μελέτη αντικτύπου εδαφικής διάστασης. Θα πρέπει επίση να διερευνηθεί η εφαρμογή και μεταφορά ε, της ε, ενωσιακής νομοθεσίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτή η πρόταση επιβεβαιώθηκε κατά τις επαφές με τα μέλη του Κοινοβουλίου, με τον κύριο Σούλτς, με τον κύριο Μπούζεκ και με την κυρία Χιούμπνερ, καθώς και με τους τρεις ε, εισηγητές της ΑΦΚΟ. Καλωσορίζω την ενισχυμένη νομοθεσία και τον ενισχυμένο πολιτικό διάλογο που έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ω Επιτροπή των Περιφερειών. Και θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή τη αρχή τη επικουρικότητα, ούτω ώστε να συμπεριλάβουμε καλύτερα ε, στην κοινοβουλευτική εργασία την Επιτροπή των Περιφερειών. Δεύτερη πρόταση. Υπάρχουν θετικά σημάδια με την πρόσφατη πρόταση προτάσεις του Συμβουλίου για το πακέτο καλύτερη νομοθεσία. Χρειαζόμαστε μια σαφέστερη αναφορά στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σχέδιο διαθεσμική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία. Να αναγνωριστεί η αναβαθμισμένη αρμοδιότητά μα που προβλέπεται από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Όμω, η καλύτερη νομοθεσία, το θεματολόγιο αυτό δεν θα πρέπει να γίνει πρόσχημα για να αποφύγουμε ή να καταργήσουμε την αναγκαία νομοθεσία. Τρίτον, επιπλέον θα μπορούσαμε να ζητήσουμε βελτίωση στις σχέσεις της Επιτροπής των Περιφερειών με το Συμβούλιο, δίδοντας ας πούμε στην Επιτροπή των Περιφερειών το καθεστώς του παρατηρητή, να μπορούμε να μιλάμε στις ομάδες εργασίας του, του Συμβουλίου σε τομεί πολιτική όπου είναι υποχρεωτικό να διαβουλευόμαστε την Επιτροπή των Περιφερειών. Παραδείγματο χάρη η δουλειά του Συμβουλίου στην πολιτική συνοχή και τι επενδύσει σε πόλει και περιφέρειες. Για πολλά χρόνια η Επιτροπή μα άκουσε το, ε, την έκκληση του πολλών κρατών μελών για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου μορφώματος του Συμβουλίου για θέματα περιφερειακά. Θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το, αυτή η έκκληση που αφορά πάνω από το 1 τρίτο του ενωσιακού προπολογισμού. Η επόμενη πρότασή μου είναι να δούμε και την προστιθέμενη αξία του να δώσουμε το καθεστώς του παρατηρητή με δικαίωμα ομιλίας στις, διαπραγματεύσει στις ε, διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου όταν υπάρχει υποχρεωτική διαβούλευση τη επιτροπή των Περιφερειών με βάση τι συνθήκε. Αυτό ήταν το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα των προτάσεων αφορά το εξή. Αν υπάρξει μεταρρύθμιση των συνθήκων, τι γίνεται. Πριν περάσουμε σε μια πιθανή αλλαγή των συνθήκων, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οποιοδήποτε αλλαγή θα πρέπει να βασίζεται σε μια ξεκάθαρη αξιολόγηση και στε... ισχυρή πολιτική υποστήριξη των κρατών μελών και των πολιτών. Θα θέλαμε να προτείνουμε κάποιες ε, προτάσεις με βάση τις συζητήσεις που είχαμε τον ε, Ιούνιο και τον Ιούλιο, στις ολομέλειες που κάναμε αυτούς τους δύο μήνες και με τα ψηφίσματα που υιοθετήσαμε πριν από μία εβδομάδα. Πρώτον, η συνθήκη της Λισαβόνας να αναγνωρίσει την αυξανόμενη σημασία των εθνικών και περιφερειών κοινοβουλίων στη νέα νομοθετική διαδικασία. Υπάρχουν νέες ναι, οι τομεί όπου η διαβούλευση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Τα μέλη μας ζήτησαν βαθμία θεσμοθέτηση της λειτουργίας της Επιτροπής των Περιφερειών ως μία δεύτερη συνέλευση, δεύτερο σώμα που γίνεται ο έλεγχος επικουρικότητας από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν θα πρέπει όμως παρόλα αυτά να αυξήσουμε τη θεσμική περιπλοκότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα δεν είναι να δημιουργήσουμε νέα θεσμικά όργανα, αλλά να βελτιώσουμε τη λειτουργία των υπαρχόντων. Να τα κάνουμε πιο πολιτικά, πιο αντιπροσωπευτικά και να λογοδοτούν περισσότερο στις πόλεις και στους πολίτες. Είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρει μια θεσμική λύση για να εξασφαλίσει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, υποχρεωτικά λένε την άποψή τους όταν διαμορφώνεται η ενωσιακή νομοθεσία που επηρεάζει τις νομικές αρμοδιότητες επιτόπου στις ε, περιφέρειες κτλ. Θέλουμε υποχρεωτικά επίσης να δίνει τη γνώμη της η Επιτροπή μας για μέτρα τα οποία επηρεάζουν τομείς πολιτικής που έχουν άμεση επίπτωση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εσωτερική αγορά, γεωργία, ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων, απελευθέρωση των υπηρεσιών, μετανάστευση, κρατικές ενισχύσεις και βιομηχανική πολιτική. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Οποιαδήποτε νομοθεσία που αφορά την εδαφική συνοχή, συγγνώμη, Πολύ σύντομα. Σας παρακαλώ γιατί έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Το τελευταίο μου σημείο. Θέλουμε μια οριζόντια ρήτρα στις συνθήκες για την ε, σταθερότητα ε, και την ε, καλή διακυβέρνηση όπου θα δίνουμε την άποψή μας για θέματα μικτής αρμοδιότητας που αφορούν το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και της νομισματικής πολιτικής. Χαιρόμαστε λοιπόν που μπορούμε να πούμε αυτές τις απόψεις και ελπίζουμε να αποτελέσουμε ε, οργανικό τμήμα της επερχόμενης διαδικασίας. Ευχαριστώ κύριε Μαρκούλα για τις προτάσεις που κάνετε για τον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο συνεισηγητές έχουν τον λόγο. Η κυρία Μερτσέντες Μπρέσκο. Ευχαριστώ. Δέκα λεπτάκια έχετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να έχουμε μεγάλη φιλοδοξία ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ότι είναι κυρίως καθήκον του Κοινοβουλίου αυτό το να κάνει ένα πολιτικό προβληματισμό για την κατάσταση της Ένωσης. Το καθήκον μας είναι περισσότερο θεσμικού χαρακτήρα. Πρέπει να προσδιορίσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να αλλάξουν αυτά που δεν λειτουργούν σήμερα. Και νομίζω ότι η έκθεσή μας θα δείξει ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο για μια τέτοια αλλαγή και αφορά και απόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα κράτη-μέλη, στην Κομισιόν, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης γενικά, κυβερνήσεις και κράτη-μέλη να κάνουν θαραλές επιλογές. Το Σεπτέμβριο που θα είμαστε και πιο πολύ άριθμοι ως Επιτροπή μπορούμε να περάσουμε στα πιο πολιτικά θέματα που συνδέονται με αυτή την περίπλοκη κατάσταση. Η εκθεσή μας προσπαθεί να μην περιοριστεί μόνο στο θέμα της ενίσχυσης της ΟΝΕ. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε βέβαια αυτό. Εξάλλου έχουμε μόλις εγκρίνει και μία έκθεση και υπάρχει και μία έκθεση επί του θέματος αυτού των πέντε προέδρων και του δικού μας προέδρου. Έτσι. Σε όλα τα θέματα αρμοδιότητας Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του χρόνου. Υπάρχει ανάγκη κατεπίγουσα, όχι μόνο στην ΟΝΕ, στην εξωτερική πολιτική, στην πολιτική ασφάλεια, μετανάστευση, άμυνας. Πολλά είναι τα κατεπίγοντα. Υπάρχουν τόσα πολλά θέματα και πρέπει να δώσουμε πολλές απαντήσεις. Πιστεύουμε πάνω απ' όλα ότι πρέπει να αναλύσουμε τη θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία και τη νομιμότητα, τη δημοκρατική νομιμότητα των θεσμικών οργάνων. Ένα από τα πρώτα σημεία επί των οποίων επί το οποίο πρέπει να προβληματιστούμε είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην ΟΝΕ, στην Ευρωζώνη, όπου από όπου προκύπτουν πολλές προτάσεις και ανησυχητικές. Δηλαδή, ad hoc κοινοβούλια, ας πούμε, που δεν θα είναι άμεσα εκλεγμένα. Δεν, μπορεί, δεν μπορούν να μας επιβάλλουν άλλες επιλογές. Θα πρέπει να συζητήσουμε για να επιλέξουμε κιόλα. Υπάρχει περιθώριο, υπάρχει δυνατότητα να στήσουμε ad hoc επιτροπές και που θα ψηφίζουν για την Ευρωζώνη. Μπορούμε να έχουμε και υπερεπιτροπές στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό της ΟΝΕ ή μάλλον και έναν υπο ε, της Ευρωζώνης δηλαδή στα πλαίσια του κοινοτικού, του ενωσιακού προϋπολογισμού. Δεν μπορώ να μακρηγορήσω σε αυτά. Αλλά όλα αυτά σημαίνουν και μία εξέλιξη δημοκρατική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μεγαλύτερη ε, χρήση της ρήτας Πασαρέλας που επιτρέπει την, νομοθετική, την τακτική νομοθετική διαδικασία για το Συμβούλιο και την ε, ψηφοφορία με πλειοψηφία στο Συμβούλιο και μία σειρά από προσπάθεια από χρήση της ενισχυμένης συνεργασίας και διαρθρωμένης συνεργασία για να βελτιωθούν οι πολιτικές. Αυτό τι σημαίνει κοινωτική μεθόδος βέβαια. Η Κομισιόν και αυτή θα μπορούσε να έχει μια δομή θεσμική μέσω της δικής της δημοσιονομικής δηλαδή ενός ε, ταμεία ας πούμε, ενός ειδικού. Η Επιτροπή των Περιφερειών, ακούσαμε τι μας ε, είπε, τι άποψη έχει και στη διαθεσμική συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να εξετάσουμε το θέμα της επικουρικότητας, οριζόντιας και κάθετης και σε υπερεθνικό επίπεδο και υποεθνικό επίπεδο που πάντα ξεκινά, ε, ξεχνάμε στις διαθεσμικές ε, συμφωνίες και το θέμα της ελεύθερης οργάνωσης της κοινωνίας που δεν θα πρέπει να καλύπτεται συνέχεια από νομοθεσία, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να οργανωθεί αυτόνομα. Σε υποεθνικό επίπεδο πρέπει να δούμε ότι αυτό το επίπεδο έχει όλο και πιο σημαντικό ρόλο εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και θα πρέπει να οριστεί καλύτερα θεσμικά. Ακούσαμε τι προτάσει, θα τι αξιολογήσουμε και θα δούμε πώ θα τι μεταφράσουμε σε κείμενο. Ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Απέναντι στο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να βελτιωθεί. Γιατί όλο και περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να εγκρίνουν ευρωπαϊκά θέματα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και θα πρέπει να βελτιώσουμε το συντονισμό μεταξύ μας. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, η οποία μας εξασφαλίζει μια σχέση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εκεί συμπεραίνουμε, καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα, σίγουρα, στα πλαίσια αυτής της σχέσης, αλλά ε, μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή τη ε, σχέση των, ε, του, του Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια μέσω των συνθηκών. Σε ό,τι αφορά την ΟΝΕ, πολλά είπαμε στις εκθέσεις που εγκρίναμε, στα κείμενα που διαθέτουμε, αλλά είναι σίγουρο ότι χρειαζόμαστε κάτι ακόμα. Πρέπει να συμπληρώσουμε την δημοκρατική πτυχή της ΟΝΕ. Υπάρχουν πολλά εργαλεία για να ενισχύσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου για να δούμε τι εκτελεστικές αρμοδιότητες έχει η Κομισιόν, για να δημιουργήσουμε εργαλεία τα οποία διευρύνουν τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης, δίνουν καταρχάς ε, στην Ευρωζώνη έναν προϋπολογισμό και υπάρχουν και κοινωνικές ε, πολιτικές ε, που υποστηρίζουν τα κράτη, τα οποία συχνά πρέπει να κάνουν επώδυνες, δύσκολες μεταρρυθμίσεις και που χρειάζονται μια κοινωνική υποστήριξη, οικονομική υποστήριξη. Έχω να πω τόσα πολλά, αλλά δεν έχω χρόνο. Φυσικά όλα αυτά τα σημεία θα τα δείτε στην έκθεση. Σημεία τα οποία μας, διευρύ, μας δίνουν τη δυνατότητα να καταστήσουν πιο δημοκρατική αλλά και πιο λειτουργική την ΩΝΕ. Συμπλήρωση επίσης της εσωτερικής αγοράς με την ε, Ενεργειακή Ένωση, με τη δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης και μιας ενίας αγοράς ε, κεφαλαίων, της Financial Union, την Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να τη συμπληρώσουμε. Είδαμε πόσο σημαντικό είναι να χωρίσουμε τον έλεγχο και την, τη διάσωση των τραπεζών από το ρόλο και τα καθήκοντα των κρατών και έχουμε και την αγορά των κεφαλαίων χρειάζεται μια δημοσιονομική ένωση. Θα πρέπει να μετασχηματίσουμε τον προπολογισμό της Ένωσης σε ένα προπολογισμό που θα βασίζεται σε ίδιους πόρους, αλλά και σε μεγαλύτερη προσπάθεια ελέγχου των φορολογικών παραδείσων, περιορισμό της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Χρειάζεται μια κοινωνική διάσταση, όπως σας είπα. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια κοινωνική ένωση που προωθεί έναν ελάχιστο μισθό, ελάχιστους κοινούς κοινωνικούς κανόνες, εναρμόνιση του συστήματος ευημερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποφεύγει το κοινωνικό ντάμπινγκ, ε, την κούσα προς τα κάτω και υποστηρίζει τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες. Τέλος. Υπάρχει και το θέμα της εξωτερικής δράσης, όπως ξέρετε. Όπως είπα πριν, στο εσωτερικό των σημερινών συνθήκων θα μπορούσαμε να φανταστούμε μία εξέλιξη προς μία πιο διευρυμένη, ενσωματωμένη εξωτερική πολιτική, καλύτερο συντονισμό και προοδευτικά μία αύξηση του ρόλου της εκπροσώπησης της Ένωσης από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο ή είπα το εκπρόσωπο που θα πρέπει να γίνει πραγματικός υπουργό εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά εργαλεία που μας επιτρέπουν να χτίσουμε μια ένωση ασφάλειας και άμυνας. Είναι οι διόψεις του ίδιου νομίσματος, δηλαδή μια κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη μετανάστευση που διαγραφήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά θεσμικά μπορεί να γίνει ε, και σε πιο ολοκληρωμένο επίπεδο. Και να δημιουργήσουμε εργαλεία για μια κοινή άμυνα. Και για ένα κοινό ναι. στρατό που θα επιτρέπει να μειώσουμε δραστικά τα έξοδα στον τομέα αυτό και να τα χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά αυτά για άλλους σκοπούς. Τελευταίο, το θέμα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Εδώ πρόσφατα είδαμε ένα προσχέδιο μιας κοινή πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που όπως είναι γνωστό πρέπει να συμπληρώσουμε και να προσχωρήσουμε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χρησιμοποιώντας καλύτερα τα εργαλεία. Αυτό όσο μπορούσα πιο γρήγορα ε, ήταν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Ευχαριστώ Μετσέντες. Θα δώσω πάρα αυτό το λόγο στον κύριο Μπρόκ. Μια και θα πρέπει να φύγει σε λίγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε το ξέρατε από πριν ότι μόνο μέχρι τις 10 μπορώ να μείνω γιατί έχουμε ψηφοφορία σε άλλη επιτροπή. 20 ή 15 λεπτά πριν την αποχώρησή μου, επιτέλους μου ζητάτε, μου επιτρέπετε να λάβω το λόγο. Ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε για διαφορετική διάρθρωση της κατανομής του χρόνου. Γι' αυτό παρακαλώ τους συναδέλφους. Ε, να σέβονται όλους τους κανόνες. Λοιπόν, δεύτερον, συμφωνούμε με πολλά από τα θέματα που ακούστηκαν, αλλά όχι επί της ουσίας. Όχι επί της ουσίας. Τίθενται θέματα ε, συνταγματικών δυνατοτήτων και η κυρία Μετσέντες ε, ε, είπε ότι πράγματι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το θέμα της πολιτικής. Νομίζω λοιπόν στο παράρτημα της έκθεσης ε, εκεί εκφράζονται διαφορετικές απόψεις και από αυτόν διεξάγεται επικοδομητικός διάλογος. Απλά ήθελα να το προτάξω αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αναφέρουμε το εξής. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μεγαλύτερη νομιμοποίηση και αυτό Και αυτό αφορά και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των ε, κείμενων ε, συνθήκων. Και αυτό δεν αφορά ε, μόνο την Ελλάδα. Να σας πω ότι θα επανέλθω επ' αυτού αλλά αφορά και στην εντύπωση την οποία γενικά προκαλεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δικαίωση αδίκως αυτή τη στιγμή αυτό δεν παίζει ρόλο. Εν πάση περιπτώσει διαπιστώνουμε ότι από πολλές πλευρές, από την άκρα δεξιά και από την άκρα, από την άκρα αριστερά, αλλά και σε άλλα στρώματα της κοινωνίας ε, αμφισβητείται η νομοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό από τελείως διαφορετικούς πολιτικούς λόγους και σκεπτικό. Άρα δηλαδή πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό έτσι ώστε να δώσουμε κάποιο μέλλον στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε οράματα αλλά και να προτείνουμε πρακτικές λύσεις, ρεαλιστικές που θα δώσουν τη δυνατότητα στους ε, πολίτες μας να κατανοήσουν ότι διεξάγεται μια διαφανής διαδικασία. Άρα δηλαδή πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν να διευρυνθούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Και εδώ ε, θεωρώ ότι πρέπει να ισχύει το, ένα αξίωμα, ε, κάτι το οποίο νομίζω το είπε, το έθιξε και η Επιτροπή των Περιφερειών. Ναι, δηλαδή το εξής, ο καθένας έχει δικαιώματα στο επίπεδο εκείνο στο οποίο έχει αρμοδιότητες. Να μην υπάρχουν κοινέ αρμοδιότητες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, δεν είναι δυνατόν να αναλαμβάνει νομοθετικές διαδικασίες. Οφείλουμε να ενισχύσουμε τα εθνικά κοινοβούλια και να δώσουμε ένα άνοιγμα έτσι ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να μπορούν να ελέγχουν και να επηρεάζουν τις κυβερνήσεις τους. Επ' αυτού υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, γιατί προφανώς αυτό υπόκειται στην στο εκάστοτε σύνταγμα, το οποίο βέβαια δεν μας αφορά εμάς καθόλου. Το τι κάνει κάθε χώρα είναι μια κυρίαρχη διαδικασία. Αλλά όχι να υπάρχει έτσι ένα αμάλγαμα που όλοι να λένε ότι υπάρχουν αποφάσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού. Αυτό είναι καθοριστική σημασία σε θέμα. Παραδείγματο χάρη, στο άρθρο 13, εκεί γίνεται λόγος ε, για το δημοσιονομικό σύμφωνο. Και εγώ θέλω να πω ότι αυτά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 13 αυτό το κοινό όργανο που έχει προβλεφτεί, αυτό το όργανο όμως δεν είναι όργανο λήψης αποφάσεων. Είναι απλά ένα όργανο όπου διεξάγονται συζητήσεις ε, και ανταλλάσσονται πληροφορίες, ακριβώς όπως συμβαίνει και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Όμως αυτό το όργανο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις, γιατί αν συμβεί αυτό τότε θα επικρατήσει πλήρης σύγχυση. Αν αυτό τώρα το μεταφέρουμε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και αυτή είναι η πρώτη που κατέθεσε ο πρόεδρος κύριος Σούλτς εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, δηλαδή στις Conversion Guidelines, εκεί να υπάρχει η δυνατότητα μέσα από μια θεσμική συμφωνία, εφόσον όλα αυτά δεν έχουν θυμιστεί στις συνθήκες, αυτές οι conversion guidelines, οι οποίες αποφασίζονται ανά πέντε χρόνια αυτές να έχουν και άμεση σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως και είναι θέμα και διοικητικό και εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παραδείγματο χάρη αν πρόκειται να κατατεθεί ένα εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων το οποίο έχει σχέση με ευρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση αυτό το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να αποφασίζεται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Άρα δηλαδή ενισχύουμε και τα δύο επίπεδα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, όχι όμως με μια πλήρη σύγχυση. Δεν θέλουμε εκχώρηση αρμοδιοτήτων, απλά οι αρμοδιότητες οι οποίες υπάρχουν να είναι δημοκρατικές και διαφανείς. Και νομίζω ότι είναι μια προσέγγιση την οποία οφείλουμε να προωθήσουμε. Κυρία Μερσέντες, συμφωνώ μαζί σας ότι πράγματι χρειαζόμαστε κονδύλια, χρήματα, για να μπορούμε να δώσουμε κίνητρα για μεταρρυθμιστικά προγράμματα. Και εδώ το πιο σωστό θα ήταν να τεθεί και το θέμα των ιδίων πόρων. Παλαιότερα, παραδείγματο χάρη, είχαμε τρία τέταρτα ίδιοι πόροι και ένα τέταρτο ε, ίδια συνεισφορά. Αυτό απέτυχε. Φτάνουμε λοιπόν λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική, σειρά, διαφορετική προσέγγιση και θα πρέπει να δούμε ανεξάρτητα αν πρόκειται για τους ίδιους πόρους ή οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να έχουμε προϋπολογισμό για την Ευρωζώνη ή για τα κράτη-μέλη τα οποία προετοιμάζονται για το ευρώ. Γιατί μπορούμε και να σκεφτούμε κατά πόσο θα πρέπει ενδεχομένω να επεκταθεί η Ευρωζώνη. Και αυτά τα οποία προβλέπονται στον κανονικό προπλησμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά είναι τα δημοσιονομικά δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως ε, μπορεί κανείς να προβλέψει κάποια κονδύλια ακριβώς για αυτή τη διαδικασία. Να πει ότι αυτά προβλέπονται για τις χώρες που προετοιμάζονται για το ευρώ. Και Τώρα έρχεται κάτι το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στο περασμένο Σαββατοκυριακό και θα παίζει πάντα ρόλο. Πρόκειται για τα προαπαιτούμενα, τα περίφημα προαπαιτούμενα. Κανεί δεν αναφέρει τα προαπαιτούμενα ή πολύ σπάνια. Δηλαδή θα προσφέρονται κίνητρα σε αυτούς που κάνουν κάτι και δεν θα είναι αυτόματες επιδοτήσει στους εθνικού προπολογισμού. Πάντα η επιδότηση θα συνδυάζεται με προαπαιτούμενα και Βεβαίως υπάρχει εδώ το περίφημο moral hazard, όσα αναφέρεται θα πρέπει να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η σκέψη θα πρέπει να ενισχυθεί, να καταστήσουμε σαφές ότι καθολής και σημασία είναι και η διάσταση της αποδοτικότητας. Έτσι λοιπόν το να υπάρχει αν θέλετε μία γερουσία των επιτροπών ή κάτι παρεμφερές, αυτό αντιβαίνει στην αρχή της αποδοτικότητας. Ε, το μόνο που πρέπει να υπάρχει είναι δύο επίπεδα, το Συμβούλιο Υπουργών και το Κοινοβούλιο. Και εκεί λοιπόν πρέπει κανείς να σκεφτεί πώς είναι δυνατόν η Επιτροπή των Περιφερειών αλλά και η ΟΚΕ κατά πόσον αυτά τα δύο όργανα μπορούν να προβληθούν περισσότερο, να συμμετέχουν περισσότερο. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές και θέματα πρακτικής φύσης... όχι θέματα αρχών. Ε, εξαρτάται βέβαια και από τους εισηγητές ε, αυτών των δύο θεσμών που προανέφερα το κατά πόσον έγκαιρα έρχονται σε επαφή με τους δικούς μας εισηγητές για να τα κουβεντιάσουμε μερικές φορές αυτό γίνεται, άλλες πάλες όχι γιατί ξέρετε κάτι πολλές φορές τη γνωμοδότηση αυτών των δύο ε, θεσμών ε, την παίρνουμε όταν ήδη έχουμε ξεκινήσει τις τροπολογίες καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί πλέον να ληφθεί υπόψη γι' αυτό λοιπόν το θέμα είναι κατά πόσον μπορούμε να προβούμε σε μια πρακτική σε συμφωνία έτσι ώστε ο δικός μας ο εισηγητής ε, να πηγαίνει στην Επιτροπή των ε, Περιφερειών έγκαιρα να συζητάει με τους ε, αρμόδιους συναδέλφους από την Επιτροπή των Περιφερειών να τους δώσουμε και χρήματα για να συναντιόνται το μεσημέρι να τρώνε αν δεν έχουν λεφτά για το μεσημεριανό γεύμα. Τι να πω κι εγώ. Θα πρέπει λοιπόν πολύ πρακτικά αυτοί οι άνθρωποι να συναντιούνται έγκαιρα μόλις ξεκινάει η νομοθετική διαδικασία να υπάρχει αυτή η συνεργασία χαριτολογώντας τα είπα όλα αυτά, φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι εννοώ, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλύτερη συνεργασία σε αυτούς τους τομείς και ε, νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το νομοθετικό μας έργο. Αυτό ισχύει για το Κοινοβούλιο, ισχύει και για το Συμβούλιο. Πρόσφατα σε μια επιτροπή της ΟΚΕ είπα ότι υπήρξα κάποτε και εισηγητής ε, της ε, Okay. Υπήρχε κάποια ε, νομοθετική διάταξη για το ωράριο ε, εργασίας ε, των οδηγών φορτηγών και εκεί διαπίστωσα ότι ούτε και στην ΟΚΕ δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι. Και τότε είπα και εγώ, ε, αφού αυτοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν, τώρα εγώ τι ρόλο έχω εδώ. Και ξέρετε τελικά τι έγινε. Προέκυψε μία ε, άποψη της ΟΚΕ και αυτή εγκρίθηκε γιατί σας είπα, επαναλαμβάνω, αν αυτοί δεν μπορούν να τα βρούνε, τι να κάνουμε. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Καταλήγοντας, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, πολύ καλύτερη συνεργασία ε, με τους θεσμούς, με την Επιτροπή των Περιφερειών και με την ε, ΟΚΕ. Να συμμετέχουν αυτοί στην νομοθετική διαδικασία και ως εκ τούτου η Επιτροπή των Περιφερειών εδώ αναλαμβάνει ιδιαίτερο ρόλο. Βεβαίω θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να καταστήσουμε σαφές ότι οι επιτροπές ε, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πολύ περισσότερο στην Ευρώπη σε αυτή την νομοθετική διαδικασία από ότι στα κράτη-μέλη. Αν δούμε λιγάκι την επιρροή που έχουν οι περιφέρειες ας πούμε στη Μεγάλη Βρετανία πραγματικά εκπλήσωμε που έρχονται εδώ οι Βρετανοί και λένε να γίνουν αυτά στην Ευρώπη, στη δική τους την πατρίδα ούτε καν να μιλήσουν δεν μπορούν. Αυτή είναι μια πρακτική. τέλο πάντων, αναφέρω, μπορώ αν θέλετε να σας πω και άλλες ε, χώρες, ακόμα και στη δική μου τη μεγάλη ομοσπονδιακή δημοκρατία, τα κρατήδια και οι ε, τοπικές ε, κυβερνήσεις, ούτε και αυτές κουβέντα δεν μπορούν να πούνε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε κατά νου. Τίθεται και το θέμα του περιεχομένου. Δεν ξέρω ε, κατά πόσον ε, ε κύρια Μεσέντη στην δική μας δουλειά να τοποθετηθούμε για τον κατώτατο εγγυημένο μισθό. Αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Ε, δεν είναι θέμα συνταγματικό. Επίσης θεωρώ ότι τα θεσμικά θέματα είναι θέματα εθνικής ε, αρμοδιότητες και εξ όσων γνωρίζω ε, σε όλα τα κρατημέλη υπάρχει ο εγγυημένος ε, κατώτατος μισθός και εν πάση που δεν υπάρχει να το λύσουν τα κράτη, δεν είναι να το ρυθμίσουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει και διαφορά στις εθνικές οικονομίες και ως εκ τούτου δεν είναι και εύκολο να εναρμονιστούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Δεν μπορεί να ρυθμιστεί το συνταξιοδοτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν η Ολλανδία και η Ρουμανία να δίνουν τις ίδιες συντάξεις. Ας το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Και πάμε τώρα στην Ελλάδα. Οι Έλληνες έχουν μέση σύνταξη που είναι ακριβώς η ίδια από αυτή των Γερμανών και διπλάσια από αυτή των Σλοβάκων. Αυτό είναι γεγονός. Εξίσου στο ίδιο ύψος η μέση σύνταξη στην Ελλάδα όπως και στη Γερμανία και διπλάσια από αυτή των Σλοβάκων. Αλλά γιατί την έχουν αυτή τη σύνταξη οι Έλληνες. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν έχουν σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μετά από ένα χρόνο ανεργίας δεν έχουν καμία απολύτως κοινωνική προστασία. Και γι' αυτό πρέπει να τους βοηθήσουμε να οικοδομήσουν ένα κοινωνικό σύστημα. Στην, ε, στην Ελλάδα όλα χρηματοδοτούνται από τη σύνταξη. Αν κάποιο είναι άνεργο, εξαρτάται απόλυτα από τη σύνταξη των γονιών και των παππούντων. Αυτό είναι το σύστημα. Αν υπάρξει μόνο μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού και καμία άλλη, τότε θα πρέπει να βοηθήσει, παραδείγματος χάνει κανείς στην Ελλάδα, να ε, θέσει επιτάπητος ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, γιατί δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα θέμα όπου μπορούμε να προσφέρουμε κίνητρα. Σχεδόν σε όλα τα κράτη υπάρχει ε, μια ελάχιστη εξασφάλιση, αλλά όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα όχι. Ακόμα και αν η Ελλάδα εισαγάγει αυτή τη σύνταξη 67 που υπάρχει ήδη σε όλα τα κράτη-μέλη, για εξηγήστε το, να πρέπει κανείς να δουλέψει στα 67, ενώ στην Ελλάδα βγαίνουν στη σύνταξη στα 50 με διπλάσια σύνταξη από ό,τι άλλες χώρες και για πέστε τώρα στο Σλοβάκο ότι πρέπει να χρηματοδοτεί στην Ελλάδα. Για πέστε το στο Σλοβάκο και στο Λετωνό. Πρέπει να σας πω ε, που δεν είδε θα να βρίσκομαι στη θέση αυτών των κυβερνήσεων ε, που θα πρέπει να θεσμοθετήσουν ρυθμίσει για να λειτουργήσει το σύστημα. Να το δείτε και από την άλλη πλευρά. Όχι να λέμε μόνο ότι αυτά τα οποία έγιναν στο Σαββατοκύριακο είναι έλλειψη αλληλεγγύης και σας το λέω αυτό κυρία Σπινέλη. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο ε, συμμετείχα σε όλη τη δικασία στο πλαίσιο των εργασιών του ΕΛΚ γιατί συμμετέχω σε, αυτή την, ε, σε αυτό, αυτές εργασίες του ΕΛΚ και διαπίστωσα ότι δεν ήταν ε, κακοί μόνο οι Γερμανοί αλλά δεν υπήρχε πια η προτιμία να συνεχιστεί η κατάσταση σε όλους, σε όλους από τη Μεσόγειο μέχρι την Ιρλανδία και τη Λετωνία. Ήθελα να τραβήξουν μία οριστική γραμμή. Τέλος πια και αυτό όχι μόνο σε κυβερνήσεις με κυβερνών κόμματα τους χριστιανοδημοκράτες. Και δεν ήταν μόνο ο κακός ο Σόιμπλε, αλλά δεν ήταν μόνο εκείνος που είχε το πρόγραμμα Α και το πρόγραμμα Β, που είχε πει ότι αν δεν περάσει το Α να περάσει το πρόγραμμα Β, το Brexit. Και όταν αυτό ελέγχθη ξεκάθαρα, έτρεξαν όλοι στο πρόγραμμα Α και προσπαθούν να βρουν ε, πλειοψηφίες στο Κοινοβούλιο. Η Ελλάδα, αν πριν από τρεις εβδομάδες είχε δεχτεί τότε το πολύ καλύτερο πρόγραμμα και δεν είχε ακολουθήσει αυτό το ε, δημοψήφισμα και οι θεατρικές ε, εξάρσεις θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα και η ευθύνη εναπόκειται καθαρά και μόνο στην ελληνική κυβέρνηση. Πριν από τρεις εβδομάδες θα μπορούσε να είχε κλείσει το θέμα αυτά είχα να πω επί της αλληλεγγύης και της ε, δημοκρατίας και τα 18 άλλα με συγχωρείτε αλλά και αυτά έχουν δημοκρατία και όχι μόνο μια χώρα η οποία διεξάγει ένα δημοψήφισμα σε λάθος χρονική στιγμή και όπου το ερώτημα του δημοψηφίσματος είναι τι θες. Θες περισσότερους ε, φόρους ε, ε, ή θες να σου περιορίσουν τις αποταμιεύσεις σου. Ε, τι να απαντήσει κανείς σε αυτό. Σας είπα λοιπόν το ποια είναι η άποψή μου και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να αλλάξουμε το κοινοβούλιο. Σας τα είπα όλα αυτά γιατί θεωρώ ότι πρέπει να τροποποιηθεί η κατάσταση και σε νομοθετικό επίπεδο. Οφείλουμε λοιπόν να καταστήσουμε σαφές ότι δεν επιθυμούμε απαραίτητα να υπάρχει ένας νέος θυσμός που να αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο ευρώ όσον αυτό που επιθυμούν ε, οι Γάλλοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει άμεση σχέση με το ευρώ και το ευρώ έχει άμεση σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όλα τα άλλα τα οποία λέγονται έχουν άμεση σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Ολάντ ας λέει ότι θέλει αλλά το να λέει ότι η πρόταση είναι να υπάρχει κοινή αρμοδιότητα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό είναι μια πρόταση που την καταποβάλλουν οι Γάλλοι ανά δύο χρόνια. Πρέπει λοιπόν να αντισταθούμε σε αυτό αν δεν θέλουμε να εγερθούν νέα τύχη στην Ευρώπη. Και εγώ δεν θέλω ως Γερμανός μια χώρα όπως η Πολωνία να ενταχθεί σε δεύτερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πολωνία βαντίζει ταχύτατα προς το ευρώ και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χώρα δεύτερης ε, κατηγορίας. Σε τελική ανάλυση νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε κάποια λύση, αλλά και εγώ πιστεύω ότι η συνθήκη το αφήνει το θέμα ανοιχτό, αυτές οι προτάσεις που υπάρχουν ε, για την Ευρωζώνη, εκεί η συνθήκη προβλέπει ξεκάθαρα ότι ο αντιπρόεδρος για θέματα οικονομικά και νομισματικά αυτόματα θα είναι και πρόεδρος της Ευρωζώνης. Και η Κομισιόν θα είναι εκείνο το εκτελεστικό όργανο το οποίο ήδη προβλέπεται και δεν χρειάζεται να υπάρχει ειδική γραμματεία για την Ευρωζώνη. Αυτά όλα έχουν ήδη προβλεφτεί. Και πρόεδρος της ε, Ευρωζώνης ε, προφανώς ε, ε, αν είναι κανείς ευφύης θα πρέπει να θεωρεί ότι είναι κάποιος που προέρχεται από το χώρο της Ευρωζώνης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα επαναλαμβάνω όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ κύριε Μπροκ. Αυτά. Καλό θα ήταν να ακούσουμε και την αντίδραση της Mercedes για το θέμα του ελάχιστου μισθού, του κατώτατου μισθού. Γιατί δεν νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό το θέμα οι δυο σας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, εισηγητές, τους κοιόδης εισηγητές. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Ο κατώτατος μισθός είναι θέμα πολιτικής αξιολόγησης και όχι συνταγματικής φύσης. Δεν είναι δική μας δουλειά εδώ να μιλάμε για τον κατώτατο μισθό. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να μιλάμε για κατώτατο μισθό, ούτε για άλλα παρεμφερή θέματα. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει εμείς να αποφασίσουμε αν θα... τι γίνεται με τον κατώτατο μισθό. Όμως υπάρχει μια κοινωνική πτυχή, ειδικά για την Ευρωζώνη, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν το συνόλο της. Και είναι αδύνατον αυτό να το λάβουμε υπόψη στο εσωτερικό των συνθήκων. Και αυτό δεν αφορά ένα ελάχιστο, ένα κατώτατο μισθό σε ευρώ, χίλια ευρώ. Έτσι. Αλλά έχει να κάνει φυσικά με, το, με τα εισοδήματα των κρατών. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε κοινού κανόνε σε κοινωνικό επίπεδο που θα ελέγχονται όπω ελέγχονται και κοινοί κανόνε σε οικονομικό επίπεδο. Γιατί γιατί το κοινωνικό dumping είναι από ένα από τα προβλήματα της εσωτερικής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια για την εσωτερική αγορά και επομένως μπορεί να έχει κανόνες που θα απαγορεύουν το κοινωνικό dumping. Αυτός είναι ο νομικός λόγος του να υπάρχει μια πτυχή κοινωνική, ειδικά για την Ευρωζώνη, που ρυθμίζεται από δημοσιονομικούς κανόνες πολύ αυστηρούς. Ευχαριστώ Μερτσέντες. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου σε αυτό το σημείο. Και τώρα, ο κύριος Ζοντόφσκι έχει το λόγο. E, e, Ευχαριστώ κύριο Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Το πρόβλημα είναι μεθοδολογικό γιατί για δεύτερη φορά μιλάμε για μια επέκταση, παράταση, χωρίς να έχουμε λάβει κανένα γραπτό κείμενο από τους εισηγητές, εκτός από την Επιτροπή των Περιφερειών και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Είναι πιο δύσκολο για μας να τα συζητήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους συνεισηγητές να ενηλικιωθούμε επιτέλους με βάση γραπτά κείμενα Αλλιώς δεν μπορούμε να συζητήσουμε μόνο με βάση προφορικές προτάσεις. Εδώ μιλάμε για την, τα μεγάλα ευρωπαϊκά ιδεώδη, για την άμυνα, αλλά πολλά από τα κράτη-μέλη δεν πληρούν τα κριτήρια ούτε και το κύριο μέλος την πατρίδα του κυρίου Μπρόκ δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στις πρακτικές ιδέες που έχουμε να συζητήσουμε. Αν θέλουμε να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία με τις εθνικές βουλές, αυτό πρέπει να γίνει με βάση κάποιον αυτοπεριορισμό. Δηλαδή, αν υπάρξει κίτρινη κάρτα, τότε να σταματάει η νομοθετική διαδικασία διότι αντίθετα από αυτά που είπε ο κύριος Μπρόκ τα εθνικά κοινοβούλια έχουν πετύχει τώρα τη δυνατότητα να μπουν και αυτά μέσα στη σφαίρα τη θεσμική σφαίρα της Ένωσης να παίξουν και αυτά ένα ρόλο δεν περιορίζονται μόνο στα καθαρά εθνικά θέματα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής των Περιφερειών να τον ρωτήσω μάλλον, εάν εννοούσε αν είχε σκοπό να υποβάλει καμία συγκεκριμένη πρόταση για να παίξει ενισχυμένο ρόλο και η Επιτροπή των Περιφερειών στη συνεργασία, ας πούμε στις πρώτες φάσεις της νομοθετικής διαδικασίας, μήπως θα έπρεπε να γίνεται κάποια συζήτηση με την Επιτροπή των Περιφερειών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με βάση της βέλτιστες πρακτικές. Δυστυχώς έχει φύγει ο κύριος Πρόμκ, αλλά είναι εδώ οι Μερθέδες. Κατά τη γνώμη της αυτές οι προτάσεις, μερικές από αυτές τις προτάσεις δεν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μια διαθεσμική συμφωνία και αν ναι, τότε θα μπορούσαν τα πράγματα να επιταχυνθούν διότι η Λουξεμβουργική Προεδρία ήδη ανακοίνωσε ότι θα ήθελε τέτοια διαδικασία να καταλήξει μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό θα ήταν θετικό για τη δουλειά μας και καλή ιδέα να, να σκουμποθούμε και να το κοιτάξουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος, ο κύριος Κόρμπετ. Ευχαριστώ. Καταρχάς για αυτά που είπατε στην αρχή κυρία Πρόεδρε. Πράγματι πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η συζήτηση για αυτά που έγιναν με την Ελλάδα να χρωματίσει την αντίληψη που έχει ο κόσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δικό μας καθήκον είναι νομίζω να μην υπεραπλοποιήσουμε αυτό το πολύπλοκο πρόβλημα και ιστορικά και ως δεδομένα και ως συμφωνία. Να δεχτούμε ότι είναι απλώς θέμα ότι η Ένωση και το Δουνουτού επέβαλαν την λιτότητα στην Ελλάδα όταν ταυτόχρονα υπάρχει μία τρίτη συμφωνία διάσωσης για την Ελλάδα μετά από ένα πρώτο κούρεμα του χρέους είναι λίγο υπεραπλουστευτικό. Χωρίς την ελάφρυνση του χρέους και χωρίς τις συμφωνίες η λιτότητα στην Ελλάδα θα ήταν ακόμα χειρότερη. Πρέπει λοιπόν να δούμε τις λεπτές αποχρώσεις του προβλήματος και να μην τα λέμε όλα απλουστευτικά. Είναι πολύπλοκο το πρόβλημα και έχει χειροτερέψει από τις ε, συνεχείς επαναχωρήσεις και διαφοροποιήσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αφού ζήτησε από το λαό να ψηφίσει όχι μετά να έρχεται και να τα δέχεται όλα και ταυτόχρονα να χάνονται εβδομάδες οικονομικής ζωής από το κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών. Λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ψέξουμε και τις δύο πλευρές. Τώρα για το θέμα του τι πρέπει να κάνουμε τώρα, τι μπορεί να γίνει με τις υπάρχουσες συνθήκες και τι απαιτεί αλλαγή των συνθήκων. Να μην υποτιμήσουμε τι μπορεί να γίνει με βάση τις ισχύουσες συνθήκες χωρίς να χρειάζονται αλλαγές. Είτε για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, που είναι μάλλον αυτό που προτιμούν οι χώρες της Ευρωζώνης, μπορούν να υπάρξει εμβάθυνση χωρίς αλλαγή των συνθήκων και απ' την άλλη τα θέματα που απαιτούν αλλαγή των συνθήκων, όπως τη συμπερίληψη των εθνικών χρεών. Εδώ όμως δεν υπάρχει συνένεση και άρα δεν θα γίνει αυτή η αλλαγή των συνθήκων. Υπάρχει όμως χώρος εμβάθυνσης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια. Δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου το εργαλείο που έχουμε για την μόνιμη συνεργασία ακόμη και αν χώρες μέλη, μερικές χώρες μέλη μπορεί να μην το θέλουν. Για τα θεσμικά επίσης μπορεί να γίνουν πολλά. Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε μια νέα διαθεσμική συμφωνία για την καλύτερη διαχείριση και νομοθεσία, καλύτερες διαδικασίες διαβούλευσης κλπ. Όπως ακριβώς στην Επιτροπή των Περιφερειών, όπου μπορούν να γίνουν περισσότερα όπως είπε και ο κύριος Μπρόκ άτυπα αλλά και επίσημα υπάρχει ε, μία μίνιμουμ διορία ενός μηνός δε μίνιμουμ θα πει ότι μπορεί να δοθεί και περισσότερος χρόνος χωρίς να χρειάζεται γι' αυτό αλλαγή των συνθήκων πολλά λοιπόν μπορούν να γίνουν και στο θεσμικό τομέα χωρίς αλλαγή το ίδιο με τα εθνικά κοινοβούλια συμφωνώ ότι πρέπει να ενδυναμωθεί η συνεργασία μας εάν κάνουν περισσότερα και οι χώρες μέλη όπως κάνουν στις βόρειες χώρες. Και αυτό δεν απαιτεί καμία αλλαγή συνθήκων. Συμφωνώ με τους εισηγητές για το διπλό ρόλο που μπορεί να παίζει η Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Ε, γι' αυτό απαιτείται απλώς ο αρμόδιος επίτροπος να έχει δύο αρμοδιότητες. Επίσης η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων δεν χρειάζεται να θεωρηθεί θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν μια ειδική γενική διεύθυνση της Κομισιόν χωρίς να είναι χωριστή η υπηρεσία ολόκληρη και για τους ιδίους πόρους εάν συμφωνήσουμε από αυτό πράγμα που είναι δύσκολο μπορεί να γίνει με τις υπάρχουσες συνθήκες η συμφωνία αυτή. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν νομίζω ότι η κύρια βελτίωση που μπορεί να γίνει αφορά καλύτερη χρήση των υπαρχουσών συνθήκων. Εφόσον μάλιστα είναι δύσκολη η αλλαγή των συνθήκων λόγω και της δύσκολης κατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου η δεξιά των συντηρητικών προσπαθεί να οθήσει τον Κάμερον σε ανεφάρμοστα αιτήματα και ζητούν πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν χωρίς αλλαγή των συνθήκων. Να το πάρουμε και αυτό υπόψη μας όταν συζητάμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη θεσμική λειτουργία της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόρμπετ. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει εντελώς το χρόνο ε, καλύψαμε όλο το χρονικό περιθώριο που είχαμε και το ξεπεράσαμε, ίσως πέω και εγώ βέβαια. Επομένως, θα είμαι πολύ αυστηρή με τους επόμενους ομιλητές. Ένα λεπτό το πολύ. Ο κύριος Φάνεμανς. Μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό θα μου δώσετε να μιλήσω γιατί είμαι εδώ από τις 9 το πρωί. Άκουσα τον κύριο Μπρόκ, την κυρία Μπρέσο και όλους τους άλλους Πρόκειται λοιπόν για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και μου δίνεται μόνο ένα λεπτό χρόνο. Τώρα δεν είναι σωστό αυτό, διαμαρτύρομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω παρόλα αυτά μέσα ένα λεπτό να σας παρουσιάσω το όραμά μου. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι κατανοείται ακριβώς ε, περί πρόκειται και τι διακυβεύεται. Στην εισαγωγή είπατε κυρία Πρόεδρε ότι θεωρείτε ότι η χρονική στιγμή είναι ακατάλληλη μετά από όλα αυτά που βιώσαμε το Σαββατοκύριακο ε, μετά το ερώτημα που έχει τεθεί τι θα γίνει ο κύριος Κόρμπετ είπε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί οποτεδήποτε πρόκειται για μεταρρυθμίσεις και διεύρυνση των ε, συνθήκων τον γνωρίζει τον κύριο Κόρμπετ, είναι ρεαλιστή, αλλά ξέρετε κάτι, αυτά βρίσκονται σε εκδιαμέτρου αντίθεση, αντίθετη κατεύθυνση προς ε, εκθέσεις που ζητούν εμβάθυνση της Ευρώπης και νέους ενδεχομένους ε, κανόνες, πλειοψηφικούς κανόνες. Ε, θα ήθελα να πω στον συνάδελφο ότι εγώ αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχω κανένα έγγραφο μπροστά μου, τίποτα το γραμμένο. Βασικά συμφωνώ με την Επιτροπή των Περιφερειών και εγώ ε, προέρχομαι από μια περιοχή, την, Φλαμαν... την Φλάνδρα, που και αυτή βέβαια πολύ ωραία θα ήταν κάποια στιγμή να γίνει ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα δούμε αυτά. Ε, αυτή τη στιγμή η Επιτροπή των Περιφερειών είναι πάρα πολύ σημαντική. Εχθές ήμουν στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και εκεί ζήτησαν όλοι τον εξευρωπαϊσμό ε, και των νομισματικών διαβουλεύσεων. Ακούγοντας λοιπόν όλα αυτά που λέγονται, είναι σαν να πρόκειται για μία περαιτέρω εμβάθυνση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, περισσότερη Ευρώπη και θεωρώ ότι λείπει ο ρεαλισμός. Στην εισαγωγή σας ε, κυρία Πρόεδρε μας είπατε και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να προχωρήσουμε ε, πιο αργά, με πιο αργό ρυθμό και να ικανοποιήσουμε βέβαια και την Επιτροπή των Περιφερειών. Γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι περισσότερη Ευρώπη αυτή τη στιγμή ίσως να μην είναι ο καλύτερος δρόμος. Κυρίως ακούγοντας πως μερικοί ζητούν ε, περισσότερες αρμοδιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία, κύριε Χάνεμανς. Η κυρία Σιλβί Γκουλάρ, ε, έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στο ένα λεπτό. Ήθελα να πω ότι είναι κρίμα που έφυγε ο Έλμερ Μπρόκ γιατί υπάρχει τρόπος να συνδυάσουμε αυτά που είπε για την ενότητα του Κοινοβουλίου και την αναγκαιότητα να υπάρξει ένα Κοινοβούλιο της Ευρωζώνης. Η σωστή λύση θα ήταν ένα Κοινοβούλιο της Ευρωζώνης μέσα στο υπάρχον Κοινοβούλιο χωρίς να δημιουργηθούν νέοι θεσμοί, χωρίς επικαλύψεις, χωρίς αποκλεισμό κανενός, απλώς να γίνονται όλες οι συζητήσεις με όλους και τη στιγμή που πρέπει να ψηφίσουμε ορισμένα πράγματα ας πούμε το ESN ή θέματα που αφορούν απλώς την Ευρωζώνη να είναι λιγότεροι συμμετέχοντες στην ψηφοφορία. Τώρα για τη Βρετανία λένε English vote for English topics, εκείνο προτείνουν. Α, μόλις απορρίφθηκε, καλά, αλλά πάντως δεν ήταν κακή ιδέα. Και το κοινοβούλιο της Βρέμης νομίζω έτσι δουλεύει. Όχι νέοι θεσμοί λοιπόν και σεβασμός φυσικά και της ενότητας και της θέλησης να μπουν και άλλες χώρες στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Mercedes. Proprio veramente uno solo. Ένα σχόλιο μόνο. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συναδέλφου που μετά το... ότι μετά το μεσημεριά... καλοκαιρινό διάλειμμα θα υπάρξει ένα έγγραφο. Ανοιχτό έγγραφο. Ούτως ώστε να ξεκαθαρίσουμε τον προσανατολισμό και την κατεύθυνση που παίρνει η Επιτροπή μας. τώρα θα πω κάτι στην Σιλβί Γκουλάχ, τα Ιταλικά, γιατί μιλάει Ιταλικά. Σίγουρα η πρόταση πάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Μια οργάνωση που μας τη ζητούν πολύ. Κοινοβούλια και κυβερνήσεις της ε, Ευρωζώνης. Αλλά που θα αφήνει όλους χώρο, σε όλους χώρο για να συμμετέχουν. Τον κύριο Κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν μέσω μιας διαθεσμικής συμφωνίας. Βασιζόμαστε στην Λουξεμβουργέζικη Προεδρία, την οποία έχουμε εδώ. Ελπίζουμε να τελεσφορήσει αυτή η διαθεσμική συμφωνία και στο εσωτερικό αυτής μπορούν να μπουν πολλά πράγματα. Ό,τι ξεφεύγει από τις συνθήκες. Και η ΕΟΚΕ και η Επιτροπή των Περιφερειών μέσω των εγγράφων τους και των συζητήσεων όπου μας κάλεσαν μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη διαθεσμική συμφωνία. Θα συμφωνήσει η Προεδρία του Λουξεμβούρου, φαντάζομαι. Ε, ευχαριστώ και συμφωνώ με τον κύριο Χάνιμαντς, με τον οποίο δεν συμφωνώ σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά σε αυτό συμφωνώ ότι ο ρόλος των υποεθνικών κυβερνήσεων, δηλαδή των τοπικών αρχών που έχουν νομοθετικό, νομοθετική εξουσία, θα πρέπει να ρυθμίζεται και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορείτε να δεν μπορούμε να ξεχνούμε εμεί ότι στο εσωτερικό των εθνικών κρατών υπάρχουν πολλά επίπεδα. Ο κύριος Κόρμπετ έκανε ω συνήθω παρατηρήσεις πολύ κέρυες. Όλα μπορούν να γίνουν αν υπάρχει πολιτική βούληση εντός των συνθήκων και κατεπηγόντω που ζητάνε πολύ. Πάντω, ε, για να αλλάξουν συνθήκε, χρειαζόμαστε πολύ χρόνο και πρέπει να πάρουμε... και χρειαζόμαστε Γρήγορε αποφάσει. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε τώρα. Σε καμία περίπτωση όμως, αν χρειαστεί, μπορεί προ το τέλο της κοινοβουλευτική μας θητεία να ανοίξει και το θέμα των συνθήκων. Δεν μας εμποδίζει κανείς. Και θα μα το πει, θα πει και την άποψή του και ο συνάδελφο Φερχόφστα. Τελευταίο ερώτημα. Θα απαντήσω σε αυτό. Για να δώσω το λόγο και στη Λουξεμβουργέζικη Προεδρία το να έχουμε μόνο ένα νομοθετικό συμβούλιο, όπως υπήρχε στη συνταγματική συνθήκη, που δεν υπάρχει σημερινή συνθήκη, αλλά δεν απαγορεύεται, έτσι. Καλό θα ήταν για, να έχουμε ένα πραγματικό ε, συνομιλητή. Θα πρέπει την οτροπία ενός νομοθετικού οργάνου να την έχει το Συμβούλιο. Εντάξει, κάποια συμβούλια συντονίζουν τις εθνικές πολιτικές, αλλά να υπάρχει ένα. Ας το διαλέξουν, το γενικό υποθέσεων ας πούμε, αν θέλουν, που πάντα ε, θα ψηφίζει με τρόπο διαφανή, ε, δημοκρατικό, με βάση ε, τους κανόνες ενός ε, ιονή κοινοβουλίου ή μιας ιονή γερουσίας. Αυτό θα μπορούσε να μπει σε μια συνθήκη. Και θα υπάρξει, θα τα γράψουμε αυτά και όλα σε κείμενο. Η συζήτηση αυτή ήταν πάρα πολύ χρήσιμη γιατί όπως καταλαβαίνετε εμείς Συζητήσαμε πάρα πολύ μεταξύ μας. Ε, δεν είναι και απλά αυτά τα θέματα. Μεταξύ μας και με άλλους, όχι μόνο μεταξύ μας. Πάντως θα τα δείτε όλα αυτά στο κείμενο που θα σας δώσουμε το Σεπτέμβριο. Ε, Πριν λοιπόν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον ε, εκπρόσωπο, τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών. Δεν έχουμε χρόνο για να σας δώσουμε δυνατότητα να μιλήσετε. Μπορούμε όμως να επικοινωνήσουμε διαφορετικά, να μας στείλετε τις απόψεις σας ε, σε γραπτή μορφή και υπάρχουν και άλλες δυνατότητες σε κάποια επόμενη συνεδρίαση. Τώρα λοιπόν καλωσορίζω τον ε, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τον κύριο Νίκολα Σμιτ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της ε, Προεδρίας του Συμβουλίου. Ο κύριος Νίκολας Σμιτ, όπως γνωρίζετε, είναι υπουργό ε, Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο πλαίσιο της Προεδρίας ε, έχει αναλάβει να διατηρεί και να καλλιεργεί τις σχέσεις με το δικό μας ε, το κοινοβούλιο. Ο κύριος ε, Σμιτ έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές υποθέσεις και διότι ήταν μόνιμος εκπρόσωπος της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον 1998 έως το 2004 και έχει συμμετάσχει στη διακυβερνητική η οποία πριν από τη συνθήκη της Νίκαιας οδήγησε στην ε, ε, συνθήκη για το μέλλον της Ευρώπης. Ένα θέμα λοιπόν ε, το οποίο θα το εξετάσει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Αυτό το θέμα έχει σχέση με τις διαθεσμικές διαβουλεύσεις για καλύτερη νομοθεσία. Και αυτή νομίζω ότι θα είναι η 12η φορά που έχουμε Προεδρία Λουξεμβούργου ε, σε μια βέβαια μακρά ιστορία ευρωπαϊκή. Ε, το Λουξεμβούργο υπήρξε επανειλημμένα ε, προεδρεύουσα χώρα στο Συμβούλιο. Μου αρέσει λοιπόν πάρα πολύ αυτό το σύνθημα που έχει επιλέξει το Λουξεμβούργο για αυτή την προεδρία που λέει «Η Ευρώπη των πολιτών». Και ελπίζω λοιπόν να υλοποιηθεί αυτή η Ευρώπη των πολιτών γιατί υπάρχει μια πολύ σημαντική κρίση αξιοπιστίας. Άρα δηλαδή θα έλεγα ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζετε είναι πολύ μεγάλη. Λίγος χρόνος στη διάθεσή σας και μεγάλη πρόκληση. Κύριε Σμιτ, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορώ να σας κρύψω ότι με μεγάλη ειδονή ήρθα, προσήλθα σήμερα εδώ στην Επιτροπή σας. Πρώτον γιατί αναφέρατε ορισμένες περιπέτειες στις οποίες συμμετείχα και τη θύμισε και ο Ριχάρδος Κόρμπετ. Πρέπει πράγματι να διαγράψω μερικά πράγματα, αλλά κυρία Πρόεδρε, αφού ήμουν συνεργάτης ενός ε, Υπουργού, όταν ο πατέρας σας έκανε την περίφημη έκθεσή του που μας οδήγησε στην ενιαία πράξη, την οποία διαπραγματευτήκαμε υπό, υπό Λουξεμβουργική τότε ήδη Προεδρία, θυμάμαι ότι είχαμε εντυπωσιαστεί όταν συναντιόμασταν από την άλλη μεριά στο κτίριο Σαρλεμάνια με τον πρόεδρο της όχι ακόμη τότε θεσμικής επιτροπής για το έγγραφο εκείνο που έφερε την υπογραφή του Αλτιέρου Σπινέλη και ακούγαμε με μεγάλη προσοχή τι μας έλεγε. Είναι κάτι που με έχει συνοδεύσει πολλά χρόνια και μέχρι το σχέδιο συντάγματος το οποίο επίσης είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες. Καμιά φορά λένε ότι τα θεσμικά θέματα, τα συνταγματικά θέματα, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις είναι για ειδικού και όχι για τους απλούς πολίτες. Κι όμως εκεί στις σχέσεις εξουσίας, στην οργάνωση των δικαιοδοσιών παίρνονται οι αποφάσεις για να δούμε αν θέλουμε μια πραγματικά δημοκρατική ένωση, μια πραγματικά διαφανή ένωση μια ένωση που όπως είπατε και εσείς δημιουργεί εμπιστοσύνη και αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα και επομένως πρέπει να εξηγήσουμε γιατί τα θεσμικά θέματα είναι τόσο σημαντικά εφόσον βρίσκονται στην καρδιά των καθηκόντων και δικαιοδοσιών που έχει η Ένωσή μας που μοναδικό σκοπό έχει την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ξέρω επίσης ότι περάσαμε μία μακρά περίοδο με πολλές μεταρρυθμίσεις συνταγματικές και ότι υπήρξαν πολλές επιτυχίες και αποτυχίες και τελικά ζητήθηκε κάποια ηρεμία, μια περίοδος ησυχίας να μην ξανανοίξουν σοβαρά θεσμικά θέματα σύντομα, αλλά απ' την άλλη όλοι έχουμε την εντύπωση, τη βαθιά εντύπωση ότι είναι κρεμή ακόμη μερικά πράγματα, unfinished business και ότι πρέπει να τα ξαναδούμε πολλά πράγματα και στις συνθήκες αλλά και σε ό,τι αφορά τα γύρω από τις συνθήκες ας πούμε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Εξάλλου νομίζω ότι και εσείς έχετε πολλές ιδέες να εκφράσετε για το πώς θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις συνθήκες πράγματα που ακόμη είναι έξω από αυτές. De, euh, από ό,τι κατάλαβα λοιπόν από όσα είπατε κάνατε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Κοινοβούλιο, για τον δημοκρατικό έλεγχο. Διότι αυτό είναι το θέμα. Πώς θα υπάρξει δημοκρατικός έλεγχος ορισμένων αποφάσεων κάτι που επί πολλά χρόνια ήταν ένα απλό σύνθημα το δημοκρατικό έλλειμμα ίσως δεν είναι απλό σύνθημα Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να δούμε πώς θα μπορούσαμε πιο αποτελεσματικά να ξανακερδίσουμε τη στήριξη, την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η Λουξεμβουργική Προεδρία, όπως είπατε ήδη, επέλεξε ως σύνθημά της μια ένωση για τους πολίτες διότι η αχίλιος πτέρνα νομίζω της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή είναι. Είναι να μην μήπως χάσουμε τους πολίτες. Μήπως δεν δέχονται φυσικό το τρόπο οι πολίτες πια την Ένωση. Πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι δεν υπάρχει σωτηρία εκτός Ένωσης. Πρέπει να πιστούν οι πολίτες από γεγονότα, από αποτελέσματα, από μεθόδους, από τρόπους διαχείρισης της Ένωσης. Για μας έχουμε καθορίσει 7 κυρίους στόχους, ας μην επισέλθω σε λεπτομέρειες γιατί έχετε ακούσει τον Πρωθυπουργό μας που παρουσίασε τα κύρια θέματα της Προεδρίας μας στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα. Γι' αυτό εγώ απλώς πολύ γρήγορα θα τα υπενθυμίσω. Οικονομία, ανάπτυξη φυσικά, πώς να αναθερμανθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Υπάρχει εδώ κάτι πολύ σημαντικό που είναι το πρόγραμμα επενδύσεων της Κομισιόν. Η απασχόληση που φυσικά είναι από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες πολλών χωρών μελών με 25 εκατομμύρια ανέργους νέους και το ξέρει και η Επιτροπή Απασχόλησης αυτό διότι όπως ξέρετε και εγώ ήμουν πρώτα υπουργό Εργασίας και Απασχόλησης να δούμε δηλαδή πώς να αναθερμανθεί και η απασχόληση ιδίως των νέων και σχετικά με αυτό ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης. Βέβαια ως Προεδρία σημειώσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον τον στόχο του τριπλού κοινωνικού αλφα. Πολύ καλό, πολύ συμμεριζόμαστε αυτή την φιλοδοξία, αλλά ήρθε πια ο καιρός να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το τριπλό κοινωνικό α, με ποιον τρόπο, πώς η κοινωνική διάσταση θα μπει στη διακυβέρνηση, στην οικονομική διακυβέρνηση και διαχείριση της Ευρώπης, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο θα γίνει άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εργασίας και θα είναι ένα από τα κύρια θέματα της ποιος είναι ο ρόλος των κοινωνικών θεμάτων στο Συμβούλιο. Είπατε ότι το Συμβούλιο είναι ενιαίο αν και υπάρχουν αφιβολίες, αλλά επειδή έχω πάει σε πολλά συμβούλια, το ξέρω κι εγώ λοιπόν, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η διακυβέρνηση αυτή και στα κοινωνικά ώστε να υπάρχει συνέπεια και συνοχή. Άλλο σημαντικό θέμα είναι οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η δικαιοσύνη, η ασφάλεια και με το, την πτυχή της μετανάστευσης η σύνδεση δικαιοσύνης και ασφάλειας και ελευθερίας, πώς θα εξισορροπηθούν όλα αυτά γιατί είναι βασικό θέμα για το κράτος δικαίου. Η Ευρώπη φυσικά είναι κράτος δικαίων και δεν είναι κράτος ακριβώς και έπειτα η εσωτερική αγορά και ό,τι αφορά τα ψηφιακά. Διότι ζούμε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη τεχνική επανάσταση που θα αλλάξει πολλά πράγματα και στην καθημερινή μας ζωή και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κράτη μας η ψηφιακή οικονομία θα αλλάξει και τις διοικητικά ήθη και τις υπηρεσίες και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και φυσικά η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει δίκτυα αλλά κυρίως να προσέξει ό,τι αφορά την επιμόρφωση των νέων στην ψηφιακή τεχνολογία εκατοντάδες χιλιάδων θέσεις απασχόλησης μπορούν από την ψηφιακή οικονομία. Ανταγωνιστικότητα λοιπόν της Ευρώπης φυσικά. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Αυτό συνδέεται και με την ψηφιακή οικονομία και με άλλους τομείς μέσα σε ένα κόσμο παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Πρέπει βέβαια με τη βοήθεια και της έρευνας να ενδυναμώσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Και τέλος, η βιώσιμη ανάπτυξη που είναι και αυτό μεγάλη πρόκληση με την προτινόμενη διάσκεψη των Παρισίων όπου η Ευρώπη θέλει να είναι πρωτοπόρος στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και όλα αυτά αφορούν και την παρουσία της Ένωσης στον κόσμο. Είμαστε πραγματικά ενεργοί σε αυτόν τον τομέα. Χαιρόμαστε για αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Βιέννη όπου η Ευρώπη έπαιξε ενεργό ρόλο στη διαπραγμάτευση με το Ιράν που κατέληξε τελικά στη συμφωνία που γνωρίζετε. Αυτά. Σας έκανα έναν πλήρη αλλά σύντομο κατάλογο των θεμάτων που, με τα οποία θέλουμε να ασχοληθούμε. Τώρα μερικά λόγια για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν ειδικά. Πρώτον, καλύτερη νομοθεσία. Όλοι συμφωνούμε νομίζω ότι η καλύτερη νομοθεσία είναι ένας στόχος που αφορά τις κύριες, τα κύρια ενδιαφέροντα του πολίτη. Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται για νομοθεσία που δεν την καταλαβαίνει μόνο οι δικηγόροι οι οποίοι κάνουν και διαφορετικές ερμηνείες. Και καμιά φορά για την ερμηνεία χρειάζεται να πάει κανείς στο δικαστήριο. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη νομοθεσία, να μην υπάρχουν νομοσχέδια όπου δεν χρειάζονται. Και εδώ λοιπόν να ισχύσει η αρχή της επικουρικότητας, ταυτόχρονα όμως να μην περικόψουμε τις δυνατότητες μας για νομοθέτηση. Πρέπει και εδώ η Ευρώπη να βρει την καταλληλότερη ισορροπία. Πού είναι σωστότερο να παρέμβει η Ευρώπη και πού δεν χρειάζεται. Γιατί οι χώρες, οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι κοινότητες θα μπορούσαν να λύσουν τα προβλήματα καλύτερα. Άλλο σημαντικό θέμα που θα αντιμετωπίσουμε είναι η συνεννόηση μεταξύ, η διαθεσμική συμφωνία γιατί μπορεί να σας φαίνεται περίεργο αλλά τελικά έτσι θα καθοριστούν οι σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και άρα και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας όλων των οργάνων και άρα είναι κάτι που ενδιαφέρει τους πολίτες διότι αν δεν συνεργάζονται σωστά και καλά τα, τα όργανα δεν ε, λειτουργεί καλά η Ευρώπη και άρα υπάρχει εκεί κάποια απώλεια. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν με στόχο να καταλήξουν μέχρι το τέλος του έτους. Εξάλλου άρχισαν ήδη με τη τα συμβολικά εγγένεια ενός Ευρωπαϊ... μιας Ευρωπαϊκής Συναυλίας. Ο κ. Φερχόφστατ που είναι ο εκπρόσωπός σας εκεί και ο κ. Τίμερμανς της Επιτροπής και εγώ από το Συμβούλιο ήδη συνεννοηθήκαμε και καθορίσαμε ένα πρόγραμμα εργασιών και θα αρχίσουμε ήδη από το Σεπτέμβριο με βάση ό,τι έχει ήδη γίνει από μια τεχνική ομάδα που ήδη άρχισε τις εργασίες της. Έπειτα, η πρωτοβουλία των πολιτών, επίσης κάτι πολύ σημαντικό, διότι βασίζεται στην θεσμική συνθήκη και μετά στη συνθήκη της Λισαβόνας και νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο δημοκρατικότητας πιο άμεσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι το κοινοβούλιο σας θέλει να βελτιώσει τη λειτουργία του συστήματος αυτού της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών και φυσικά το Συμβούλιο είναι έτοιμο και διατεθειμένο να το στηρίξει αυτό. Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις στο Συμβούλιο για να δούμε πού πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, τι πρέπει να βελτιωθεί και επ' αυτού νομίζω πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό, είναι θέμα ρεαλισμού. Για να δούμε δηλαδή πώς πιο αποτελεσματικά θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την λειτουργία από τεχνική αυτού του συστήματος. Κάτι τώρα για το δικαίωμα έρευνας και εξέτασης. Γιατί νομίζω ότι θα με ρωτήσετε πολύ για αυτό το θέμα. Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό διότι φρονούμε ότι το δικαίωμα αυτό αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της λειτουργίας ενός κοινοβουλίου, άρα και του Ευρωπαϊκού και προβλέπεται και από τις συνθήκες. Επομένως το Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να ασκήσει αυτό το, το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 226. Είναι θέμα δημοκρατικού ελέγχου. Το δικαίωμα λοιπόν αυτό του Κοινοβουλίου αναγνωρίζεται καθολικά ως ένα, μία από τις βασικότερες δικαιοδοσίες του πολιτικού ελέγχου και γι' αυτό το λόγο οι συνθήκες δίνουν αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κανονισμός που θα προκύψει από αυτό θα καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους θα ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και θα καθορίζει και προς ποιον θα γίνεται ο έλεγχος, απευθύνεται ο έλεγχος. Αυτό είναι νομίζω το λεπτότερο θέμα. Φυσικά οι θέσει των μελών του Συμβουλίου μπορεί να μην ταυτίζονται απόλυτα με τις θέσεις που μέχρι τώρα έχουν εκφραστεί από το κοινοβούλιο σας. Βεβαίως έχουμε πάρει, κάνει νομικές νομοδοτήσεις από την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα διότι είναι τμήμα του πολύ σημαντικού θέματος αυτό που αφορά το κοινοβουλίο σας. Τέλος, η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου, του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Νόμου. Ήδη με την πρόεδρο κυρία Χούμπνερ και τον κύριο Λάινεν κάναμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας. Προετοιμάζεται νομίζω έκθεση πρωτοβουλίας, ιδίας πρωτοβουλίας για αυτό το θέμα, η οποία δεν έχει ακόμη εγκριθεί από εσά, από την Επιτροπή σας. Φυσικά είμαστε διατεθειμένοι να παραμείνουμε σε επαφή με την Επιτροπή σας για αυτό το θέμα που δεν σας το κρύβω, είναι πολύ λεπτό γιατί αφορά και τις εθνικές δικαιοδοσίες και εκλογικά δικαιώματα. Ως Προεδρία όμως θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε από αυτού και ότι πρέπει και πάλι εδώ να είμαστε ρεαλιστές. Τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να βελτιωθεί πραγματικά για το Ευρωπαϊκό Εκλογικό Σύστημα τι λύνει τις διοικητικές, τους διοικητικούς παραλογισμούς, ας πούμε υπερβολικά μικρές διορίες και που δεν μπορούμε να τα δεχτούμε από τους εσωτερικούς εκλογικούς μας νόμους και παρόλα αυτά ισχύει για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά και η Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να προχωρήσουν και εδώ τα πράγματα. Να, αυτά ήθελα να σας πω προκαταρκτικά και σας ξανά ευχαριστώ που με καλέσατε στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ο κ. Γιολάινεν. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Είμαστε γείτονε, κάναμε πάρα πολλά μαζί. Σε αυτή τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή περιφέρεια. Χαίρομαι λοιπόν που ένας τόσο ικανός άνθρωπος αναλαμβάνει την Προεδρία. Στην ενιαία πράξη πολεμήσαμε μαζί. Έχετε μεγάλη εμπειρία. Και θα είσαστε χρήσιμος σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπιστοσύνη είναι το θέμα των τελευταίων εβδομάδων. Τις τελευταίες ε, ημέρες νομίζω κλειδονίστηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και στους πολιτικούς συθήνοντες. Γιατί η Ευρώπη είναι μια παρτίδα πόκερ. Δεν είναι μια κοινότητα ευθυνών για όλους. Στα πλαίσια ενός κοινού καλού, αλλά είναι η σκηνή όπου παίζουμε ένα πόκερ με ψέματα για το κοινό, κατά του κοινού και νομίζω ότι αυτή είναι μια απειλή που μπορεί να μας διαλύσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, να προτάξουμε το κοινό συμφέρον. Δυστυχώς υπάρχει μια τάση επανεθνικοποίησης. Θέσατε το εξής ερώτημα. Με ποιο τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε την Ευρώπη και να της αφήσουμε δημοκρατικό περιθώριο. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία ότι επανερχόμαστε στους εθνικισμούς. Επανερχόμαστε στα δημοψηφίσματα. Το επερχόμενο δημοψήφισμα στην ε, Μεγάλη Βρετανία και στη Φιλανδία δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση. Όμορφο είναι, αλλά δεν είναι η καλύτερη λύση. Γιατί μια, ένα εθνικό δημοψήφισμα για μια ευρωπαϊκή απόφαση στην πραγματικότητα είναι μια αντίθεση σε όλους τους υπόλοιπους εταίρους. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη δημοκρατία να αναπτυχθεί, να αναπνεύσει, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τη δημοκρατική Ευρώπη. Και η λέξη κλειδί είναι οι εκλογές, οι ευρωπαϊκές εκλογές για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και χαίρομαι που η Λουξεμβουργέζικη Προεδρία είναι υπέρ της ε, βελτίωσης ε, των ευρωεκλογών γιατί από, τις πρώτες, ε, από την πρώτη φορά που διενεργήθηκαν ευρωπαϊκέ, εκλογές δεν άλλαξε τίποτα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πιο ελκυστικέ οι ευρωπαϊκές εκλογές, ε, πιο αξιόπιστε, πιο σωστά διοργανωμένε. Μιλήσατε για αυτό το λεπτό θέμα. Σίγουρα το Συμβούλιο Υπουργών θεωρεί ότι οι ευρωεκλογέ είναι κάτι πολύ κακό. Φρίκι για αυτούς και επίσης μια έκθεση πρωτοβουλία για τις ευρωεκλογέ. Τι θα πούμε σε αυτή την έκθεση. Αλλά έχω εμπιστοσύνη σε εσά ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα κάνετε σημαντικά βήματα για αυτό το θέμα. Θα ήθελα επίσης να πω δύο λόγια για ένα άλλο σημείο. Είσαστε Υπουργό Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εάν έχουμε μια Ευρώπη του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας, δεν θα έχουμε καθόλου ε, τίποτα το κοινωνικό εκεί. Δεν θα υπάρχει κοινωνικό συστός. Ε, από το better regulation θα πάμε στο no regulation. Από την καλύτερη νομοθεσία δεν θα έχουμε καθόλου νομοθεσία για την κοινωνική Ευρώπη. Εάν η νομοθεσία εξυπηρετεί μόνο την Ευρώπη του ανταγωνισμού, νομίζω ότι έχουμε ακολουθήσει λάθος άγουσα. Θα πρέπει εσείς να επαγρυπνέατε, ούτω ώστε να μην ξεχάσουμε εντελώ την ε, κοινωνική διάσταση. <laughs> Σα ευχαριστώ. Όλα αυτά τα θέματα Γιολάινεν έχουν να κάνουν με την κοινωνική, που έχουν να κάνουν με την κοινωνική διάσταση, συνδέονται με τον κατώτατο μισθό και είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα κατά την άποψή μου. Η κυρία το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνική, γιατί ο κύριος Σμιτ ήταν πάρα πολύ σαφής και νομίζω ότι όλοι μας εδώ καταλάβαμε ότι με την Προεδρία του Συμβουλίου έχουμε έναν άνθρωπο φίλο της Ευρώπης, πεπισμένο ευρωπαϊστή που ξέρει και τα θέματά του. Σπάνιο είδος, εποφεληθείτε. Γιατί τους επόμενους έξι μήνες με τον Νίκο Σμιτ μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί έχει και επιθυμία να προχωρήσουμε. Το ξέρω εδώ και χρόνια. Τα έχει σκεφτεί τα θέματα, έχει λύσεις, έχει το κουράγιο να πιέσει τα πράγματα για να υλοποιηθούν οι λύσεις. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε για κάποια θέματα, τώρα είναι η στιγμή. Είναι και η ώρα γιατί έχουμε ένα σύμμαχο. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Ζοντόφσκι. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Για το... τη νέα... Η Προεδρία θα παρουσιάσει νέους μηχανισμούς, νέες ε, συγκεκριμένες προτάσεις. Δηλαδή, μια πιο αποτελεσματική νομοθεσία, ενίσχυση της αρχής επικουρικότητας. Εάν ναι, τι προτάσεις ακριβώς θα κάνει η Προεδρία. ευχαριστώ. Ο κύριος Durand. Merci, euh, Madame euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που κάνετε αυτή την παρουσίαση. Ένα αστιάκι, αν μου επιτρέπετε. Μας είπατε ότι ο θεσμικό διάλογος έχει ξεκινήσει και ότι έγιναν οι πρώτες ε, συνεδριάσει κυρίως με τον κύριο Φερχόφστατ. Ε, περίεργο σημαίνει να μάθω ποια είναι η θέση που υπερασπίστηκε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί έχει μία αποστολή ο κ. Φερχόφστατ, αλλά δεν έχουμε ούτε εντολή, ούτε μα είπε και τίποτα. Μπορείτε να μα πείτε τίποτα, έτσι, δύο λόγια. Τέλο πάντων, ό,τι θέλετε για την ερώτησή μου. Φυσικά όλα αυτά τα λέω χωρί ίχνο πολεμοχαρού διάθεση. Ε, το θέμα τη εντολή, τη προσωπευτικότητα. Ε, δεν σα αφορούν όλα αυτά άμεσα, αλλά υποφελούμε από την ευκαιρία που έχουμε εδώ να σα έχουμε μεταξύ μα, να μου απαντήσετε. Κάτι που με ανησυχεί τώρα στο πρόγραμμα εργασία. είναι αυτό το θέμα των μελετών αντικτύπου. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να υπάρχει καλύτερη νομοθεσία. Το καταλαβαίνω. Αλλά μιλάμε πολύ για τη δημοκρατία και το δημοκρατικό θέμα. Είμαι παλιός έτσι νομομαθής. Αν... Ανησυχώ που πριν ληφθούν α, αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο, στην πραγματικότητα τους επιβάλλουμε μία θεώρηση για τα πράγματα. Αυτό για τις ε, μελέτες αντίκτυπου. Κάτι το οποίο επανέρχεται κάθε φορά. Το αρχείο, το μητρό μάλλον τον λόμπι για το Συμβούλιο. Το λέω κάθε φορά. Ακούραστα. Και κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι κάποια μέρα όπως υπάρχει η διαφάνεια στη συζητήση του Κοινοβουλίου, κάποια καλή ημέρα θα έχουμε τα πρακτικά του τι διαμείδεται στο Συμβούλιο, καλό θα ήταν. υπάρχει ένας παραλληλισμό. να ξέρουμε και εμείς τι λένε αυτοί οι άνθρωποι και πώς το λένε, όπως ξέρουν και τι λέμε εμείς. Δύσκολο είναι και αυτό το ξέρω, αλλά δεν βλάπτει να θέσω το ερώτημα. Ευχαριστώ. Πασκάλ. Και εγώ θα ήθελα να μάθω. Τι σας λέει ο κύριος Φερχόφστατ. Ο συνάδελφός μας θα έρθει εδώ στις 21 Σεπτεμβρίου. Αλλά και εγώ είμαι περίεργη να μάθω τι σας λέει αυτός ο άνθρωπος στην κυρία Μπρέσο. Μετσέντες. Ευχαριστώ. Ε, ε, Καλώ ήρθατε κύριε Σμιτ. Και εμεί είμαστε πεπισμένοι ότι με τη Λουξεμβουργιάζικη Προεδρία θα προχωρήσουμε. Στα θέματα που απασχολούν την Ένωση εν το συνόλο της αυτή τη στιγμή αλλά και τα θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα στην Επιτροπή μας. Για το γενικό πρόγραμμα της ε, Προεδρίας σας, εμείς στεκόμαστε σε κάποια ιδιαίτερα σημεία. Η θεσμική οργάνωση, διοργάνωση, οργάνωση, η δομή της ΟΝΕ, ναι, ο ρόλος του Κοινοβουλίου εκεί, στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Σε μια προηγούμενη έκθεση είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα. Η συζήτηση γίνεται πολύ έντονη και μπορεί να γίνουμε ένα κοινοβούλιο δεύτερης κατηγορίας. Ε, όπως ήμασταν πριν από 50 χρόνια ένα κοινοβούλιο διορισμένο από τα κράτη. Επικεντρώστε παρακαλώ την ε, δημοκρατική σας προσοχή σε αυτό το θέμα. Είναι ένα από τα θέματα επί των οποίων θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Για να δούμε πώς παίζει το ρόλο του, πώς κάνει το δημοκρατικό έλεγχο το Κοινοβούλιο για θέματα που αφορούν την επικουρικότητα και που οδηγούν σε λήψη αποφάσεων που εκφεύγουν το δημοκρατικό ελέγχου του Κοινοβουλίου. Το είπα και το ξαναλέω. Χρειαζόμαστε περισσότερη δόση από την κοινοτική μέθοδο. Λόγω κρίσης διολυστήσαμε, την ξεχάσαμε αυτή τη μέθοδο. Και με υπομονή μπορούμε να επανέλθουμε στον δρόμο της αρετής, που είναι η κοινωτική μέθοδος. Το δεύτερο θέμα. Την τριπλή κοινωνική διάσταση. Και εδώ υπάρχουν θεσμικά θέματα. Τα κοινωνικά θέματα ανήκουν 100% στην εσωτερική αγορά γιατί κοινοί κανόνες για το welfare είναι κοινοί κανόνες. Εγώ δεν θέλω να έχουμε τον ίδιο κατώτατο μισθό όλοι σε απόλυτες τιμές, αλλά τους ίδιους κανόνες όλοι, ούτω ώστε να αποφύγουμε το κοινωνικό dumping. Και εδώ θέλω να μας πείτε πώς ορίζεται αυτό το τριπλό κοινωνικό α. Αυτή την τριπλή βαθμολογία, αυτή τη βαθμολογία α για τα κοινωνικά που το είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν. Για το, αυτό, για το έθνομοθετήν. Θέμα είναι εξελίξη. Καλό θα ήταν να μας παρουσιάσει την θέση του ο κ. Φερχόφστατ. Κάνα πρόβλημα γιατί είναι και τη Επιτροπής. Μπορούμε να το ζητήσουμε να μας πει τι γνώμη έχει. Πολύ συχνά ξεχνάμε κάποια πράγματα. Εγώ είμαι οικονομολόγος και έχω μάθει πολλά νομικά. Αλλά μου, α, είπανε ότι ο κανόνας, ο νόμος μάλλον πρέπει να είναι γενικός και ε, Αφηρημένος, αόριστος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πέρα από τα εθνικά κοινοβούλια υπάρχουν και τα περιφερειακά κοινοβούλια που μερικές φορές παρεμβαίνουν. Και το να κρατήσουμε αυτόν τον κανόνα του δικαίου που είναι ε, γενικό και αφηρημένο είναι τμήμα του εθνομοθετή. Γιατί ε, προσαρμοζόμαστε με αυτόν τον τρόπο στις διαφορετικές πραγματικότητες, της εθνικές και υποεθνικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη μας μίλησαν γι' αυτό. Βελτιώνουμε την πρωτοβουλία των πολιτών αυτή τη στιγμή. Ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Ασχολούμαστε με το δικαίωμα σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ο κύριος Ραμόν Χαουρέγγι θα μιλήσει για αυτό το θέμα και θα μιλήσουμε και για τον εκλογικό νόμο. Πολύ ενδιαφέρον θέμα και αυτό και θα θέλαμε να ακούσουμε τη θέση του Συμβουλίου γι' αυτό. Έχουμε προχωρήσει αρκετά στα κείμενα. Έχετε τη δυνατότητα. Μας πείτε τι θεωρείτε αποδεκτό και λογικό. Ένα κοινό κατόφλι, Φερρυπίν. Σαφέστερη υποχρέωση εναλλαγής των φύλων Και αυτόν το εγγυάται την νομοθεσία. Και άλλα πράγματα, όπως αυτά που είπε ο κύριος Λάινεν. Θα μπορούσε να είναι τμήμα της ε, σοδιάς που θα μας εξασφαλίσει η Προεδρία σας. Και χάρη σε αυτή θα μπορούσαμε να έχουμε μία πιο δυνατή και δημοκρατική ένωση. Βεβαίω δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε αυτά στο εξάμεινο τη Προεδρία σα με τροποποίηση των συνθήκων, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα αν υπάρχει καλή θέληση από τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα. Ευχαριστούμε πολύ, Mercedes. Θέλω να σας παρακαλέσω κάτι. Να μιλάτε παρακαλώ σύντομα. Γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουν να μιλήσουν οι υπόλοιποι και να ακουστούν και οι απαντήσεις του Υπουργού. Σας παρακαλώ. Κύριος Καστάλντο, ορίστε Φάμπιε. Σε ευχαριστώ Βαρβάρα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Είναι ευχάριστο που γίνεται αυτή η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων. Θέλω και εγώ να γραφτώ στη λέσχη των συναδέλφων που ελπίζουν σε λίγο να μιλήσουν, να συνομιλήσουν με τον κύριο Φερχόφστατ τον Σεπτέμβριο, πριν λήξουν οι διαπραγματεύσεις, εν καιρό δηλαδή. Για τις διαπραγματεύσεις λοιπόν και τη διαθεσμική συμφωνία. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της προάσπισης των δικαιωμάτων μικρών κοινοβουλευτικών ομάδων, το δικαίωμά τους έκφρασης δηλαδή, θέσης γιατί πολλές φορές είχα την εντύπωση ότι δεν του δίνουμε σημασία αυτού του θέματος. Ιδίως για τους τριμερείς διαλόγους που είναι άρνηση της κανονικής διαδικασίας που προβλέπουν οι συνθήκες. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, τι φρονείτε κι εσείς. Δεύτερον, ήξατε το θέμα της πρωτοβουλία των πολιτών. Κάτι πολύ καλό, πολύ θετικό. Μια νομική ιδέα και καθεστώς το οποίο εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα όπως και άλλους. Αλλά επίσης για το ίδιο θέμα οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν συχνά το αίσθημα ότι τους αγνοούν. Υπάρχουν πολλοί φραγμοί και δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση της Κομισιόν να απαντήσει και ακόμα περισσότερο, ακόμα λιγότερο μάλλον να αντιδράσει για τα θέματα που θα έχουν θίξει οι πολίτες. Στα πλαίσια λοιπόν ακριβώς του διαλόγου για την πρωτοβουλία των πολιτών θα ήθελα να μου πείτε Ποια είναι η θέση σας ως προς την αντίδραση που πρέπει να έχει η Κομισιόν μπροστά σε τέτοια απευθείας έκφραση της θέλησης των πολιτών. Για τον εκλογικό νόμο θα ήθελα να ξέρω τι είναι ρεαλιστικό για σας, τι εννοείτε όταν λέτε ρεαλιστική προσέγγιση. Αυτή την έκφραση χρησιμοποιήσατε. Ο αγαπητό μου συνάδελφο Διουράν είπε πριν από μένα αυτό που ήθελα να πω για περισσότερη διαφάνεια των εργασιών του Συμβουλίου. Υποστηρίζω αυτά που είπε και τέλος η ερώτηση των ερωτήσεων. Λόγω της δύσκολης περίοδου που αντιμετωπίζουμε θα ήθελα να γνωρίζω ποια αποτίμηση κάνετε των τελευταίων γεγονότων με τη Συμφωνία Δανειστών και Ελλάδος. Και εγώ είμαι πεπισμένος ότι έχουμε μια μεγάλη επιλογή μπροστά μας η οποία πρέπει να γίνει τώρα, όχι σε δύο-τρία χρόνια. Είτε θέλουμε όντως να οικοδομήσουμε μια σε εισαγωγικά ομοσπονδιακή Ευρώπη με τον ανάλογο προϋπολογισμό με πιο επεκτεταμένες οικονομικές πολιτικές και αποφυγή των φορολογικών παραδείσεων καθώς και του φορολογικού ανταγωνισμού είτε θέλουμε επίσης κάποιον επιμερισμό των κρατικών χρεών για να πραγματοποιηθεί επιτέλους αυτή η περίφημη κοινωνική ένωση του τριπλού κοινωνικού α για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργό σας. Είτε απ' την άλλη η Ευρωζώνη θα διαλυθεί από μόνη της διότι δεν πιστεύω προσωπικά ότι μπορεί να διατηρηθεί χωρίς αυτά τα εργαλεία που ανέφερα διότι οι ασυμμετρίες που παρατηρούμε σήμερα και οι επιπτώσεις τους δεν μπορούν πια να γίνουν δεκτές αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εσεί τι φρονείτε. Και προσωπικά και τι φρονεί η Λουξεμβουργική Προεδρία. Τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να κινηθούμε προς μια άλλη κατεύθυνση τους επόμενους έξι μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς ε, κύριε Καστάλντο και ακριβώς και διότι θίξατε και εσείς το θέμα με το οποίο εγώ άνοιξα αυτή τη συνεδρίαση. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Χαουρέγγιτς. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ που εμφανιστήκατε μπροστά μας, που ήρθατε στην ε, Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε, που μας μιλήσατε. Υπάρχει ένα θέμα που αναφέρατε, η σχέση ή μάλλον ε, το θέμα του, της σύστασης εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, Υπουργέ. Εσείς κάνετε τόσα καλά, τόσες καλές προβλέψεις, έτσι αισιόδοξε. Τους τελευταίους έξι μήνες θα σας πω όμως ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας και εγώ προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με το Συμβούλιο, ήταν αδύνατον. Γιατί, γιατί το Συμβούλιο, κατά τη γνώμη μου, έχει μια στάση έχθας στην, απέναντι στην έκθεση που είχε περάσει από το προηγούμενο κοινοβούλιο. Και το καταλαβαίνω. Γιατί το κοινοβούλιο δεν μπορεί να περάσει ένα νόμο με δικαίωμα πρωτοβουλία. Το μοναδικό νόμο που μπορούμε να εγκρίνουμε με κοινοβουλευτική έγκριση, ε, δεν μπορούμε το, να το κάνουμε αν δεν έχουμε και την έγκριση του Συμβουλίου. Το καταλαβαίνω. Αλλά το παλιό κοινοβούλιο, ε, για να μην πέσει στις καλένδες αυτό το θέμα, να μην περάσει στις καλένδες, το ενέκρινε. Υπάρχει τέλος, πάντως, υπάρχει τέλος πάντων αυτή η έκθεση που έχει περάσει από το προηγούμενο κοινοβούλιο και που την αντιμετωπίζει με έξτρα το Συμβούλιο. Εμείς, <coughs> εμάς μας κληροδοτήθηκε αυτή η έκθεση. Εγώ έκανα μία έκθεση πάνω σε αυτή την, σε αυτή την απόφαση και ζήτησα από τους συντρόφους της Επιτροπής να δείξουμε ευελιξία για να ε, βρούμε να εξασφαλίσουμε μια νέα συμφωνία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Προσπάθησε επί έξι μήνες να μιλήσω μαζί τους. Και η Προεδρία της Λετωνία έκανε μια τεράστια προσπάθεια. Αλλά υπήρχε μια ε, μειοψηφία ανάσχεσης στο Συμβούλιο. Και το λέω, θα πρέπει να του το πω. Και εγώ το λέω και εδώ και το λέω και σε εσά, Υπουργέ. Γιατί συγκαλέσαμε στι 18 Ιουνίου μία συνεδρίαση η οποία ακυρώθηκε από το Συμβούλιο στι 9 το βράδυ την προηγούμενη. Δηλαδή την ακύρωσαν τελευταία στιγμή. Έχω τεράστια απογοήτευση. Μάθετε ότι το Κοινοβούλιο θέλει να διαπραγματευτεί τη συμφωνία. Θέλει να υπάρξει μια ε, συνένεση μαζί σας και με την ε, Επιτροπή, γιατί έχουμε συνείδηση, έχουμε συνέστηση ότι ή θα συμφωνήσουμε είτε θα έχουμε δικαίωμα να συστήσουμε Εκταστική επιτροπή. Εντάξει. Τελευταίο και τελειώνω, Πρόεδρε. Σας ζητώ μόνο το Συμβούλιο να αρχίσει να μιλάει μαζί μας. Έκανε, έγινε μία συνεδρίαση με την Κομισιόν και ζήτησα η Προεδρία να είναι παρατηρήτρια, γιατί το Συμβούλιο δεν της έδωσε το OK για να συμμετάσχει σε μια προκαταρτική, τεχνική και άτυπη επιτροπή. Δεν της έδωσε το Συμβούλιο της Δετανικής Προεδρίας το OK, έτσι. Σας λέω με ποιο πνεύμα μιλάω. Ε, σα λέω ποια ήταν η πρόθεσή μου. Σα ζητάω απλώ να συνεχίσετε την προσπάθεια, ούτω ώστε το Σεπτέμβριο να, μπορούσα, να μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε, απλώ να μιλάμε Υπουργέ. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εγκρίνει ένα κανονισμό με τη συμφωνία σα, με τη συμφωνία, σύμφωνη γνώμη τη Κομισιόν, ούτω ώστε να υπάρξει ένα κανονισμό, ένα νόμο, ούτω ώστε να ασκήσουμε ένα δικαίωμα που είπατε εσείς ότι είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει μια τέτοια μακρά ε, κοινοβουλευτική παράδοση. Ευχαριστώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Χαουρέγγι για την τόσο σημαντική ερώτηση που υποβάλατε. Ο κύριος Σότς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ θα μπω λιγάκι βία στη συζήτηση. Και σας το λέω αυτό με ειλικρίνεια, γιατί πριν από έξι χρόνια, όταν εγώ πρωτοήρθα στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχα αρχίσει τότε να δουλεύω στη Συνταγματική Επιτροπή, μιλάγαμε για τη δημοκρατία, για την κοινωνική Ευρώπη, για τις προκλήσεις, για την κοινοτική μέθοδο, εκλογικό δικαίωμα, δικαιώματα και πρωτοβουλίες πρωτοβουλών. Κατορθώσαμε να επιτύχουμε κάποια πράγματα. Παρόλα αυτά όμως, παραμένουν όλα στάσιμα και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μεταρρύθμιση της συνθήκης. Γιατί όσο ε, έχει τώρα η συνθήκη της Λισαβόνας δεν λειτουργεί σωστά. Υπάρχουν αμέτρητες κοινωνικές και οικονομικές ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να προχωρήσουν έτσι τα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη κόποση για την Ευρώπη και στα 28 κράτη-μέλη. Ο Guardian εχθές δημοσίευσε ένα άρθρο όπου αναφέρει η αριστερά και ξέρετε τι λέει η αριστερά ο Guardian, εννοεί το εργατικό κόμμα, όχι την άλλη αριστερά. Η αριστερά λοιπόν, λέει ο Guardian, θα πρέπει να θέσει το θέμα της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάει για Lexit. Υπάρχει Grexit, Brexit. Υπάρχουν όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, όλα αυτά μπαίνουν σε πολιτικό και κομματικό επίπεδο. Εγώ σας το λέω ξεκάθαρα, είμαι κατά αυτής της στρατηγικής. Οφείλουμε να ενισχύσουμε τη διαδικασία ολοκλήρωσης, αν αντιερωτηθούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Ποια είναι η κοινωνική Ευρώπη. Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν πια στην καθημερινότητά τους να βλέπουν την Ευρώπη και διαπιστώνουν ότι αποκλείονται από τις διαδικασίες λήψη αποφάσεων και καταλήγουν στο ότι ανεξάρτητα αν τα ψηφίσουν συντηρητικούς, ελεύθερου ή αριστερούς, τίποτα πια δεν γίνεται. Ε, σε αυτό το σημείο έχουμε πια αποτύχει και νομίζω αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζει το Λουξεμβούργο, η Προεδρία του Λουξεμβούργου. Συμφωνώ με τον κύριο Καστάλντο, δεν έχουμε πια χρόνο για να παρηγοριόμαστε και γι' αυτό σας είπα ότι εγώ ξεκίνησα πριν από έξι χρόνια. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε, ε, που είπατε ότι θέλετε να θίξετε την εκλογική μεταρρύθμιση ε, της πρωτοβουλίας ε, πολιτών, την καλύτερη νομοθεσία. Τι είναι όμως αυτή η καλύτερη νομοθεσία. Με αυτήν βαντίζουμε προς την κατεύθυνση της κοινωνικής Ευρώπης ή όχι. Ή για να το πω αλλιώς, το κομβικό σημείο που δεν έχει απαντηθεί. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει εταιρική σχέση, ουσιαστική σχέση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το ε, Συμβούλιο. Δεν υπάρχει συνεργασία στο ίδιο επίπεδο. Αυτή κατ' ουσίαν είναι και η αντίφαση που υπάρχει πίσω από την κοινοτική μέθοδο και τη διακυβερνητική μέθοδο. Και αν δεν ενισχύσουμε την κοινοτική μέθοδο θα υπάρχουν όλο και περισσότερο τάσεις ε, εθνικών ε, εξάρσεων. Αυτά τα οποία έγιναν το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε. Να δούμε λιγάκι τι έγινε και τότε με τη Ιουγκοσλαβία, με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Κανείς δεν πίστευε ότι λίγους μόνο μήνες μετά τη διάλυση της ε, Ιουγκοσλαβίας θα προέκυπτε πόλεμος. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση αν μας πάρουμε σοβαρά και σκεφτούμε τι κάνουμε μόνο τότε ε, θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Και γι' αυτό λοιπόν σας λέω αυτή η Επιτροπή όπως επίσης και η οικονομική και νομισματική πολιτική του Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο στην ολομέλειά του είπε το 2014 ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτό το μόρφωμα που λέγεται Τρόικα και για συνταγματικούς λόγους. Και τι έγινε μετά, τίποτα, απολύτως τίποτα. Και σήμερα απλά διώνουμε τη συνέχιση της αποτυχίας αυτού του μορφώματος. Πιστεύω ότι και για καθαρά πρακτικούς δημοκρατικούς λόγους, όχι μόνο θεωρητικούς, οφείλουμε να βελτιωθούμε και να αντιμετωπίσουμε τα κέρια θέματα με μεγαλύτερο θάρρος. Και τελικά γιατί δεν επιδεικνύουμε θάρρος, για λόγους κομματικοπολιτικούς, για λόγους ισορροπίας εξουσιών, ίσως ε, γιατί ε, για εθνικούς λόγους ε, θέλουμε να εξασφαλιστούμε πίσω από την διακυβέρνηση. Μπας περιπτώσει, σας ευχαριστώ θερμά σήμερα για όλα αυτά που μας είπατε και ελπίζω στον απολογισμό μετά από έξι μήνες να, έχουμε, να επιδείξουμε κάτι καλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Χέλμουτ, για τις ε, θεμελιώδεις ερωτήσεις που έθεσες. Η Σιλβή Γκουλάρ έχει το λόγο. Euh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έχω ένα μήνυμα μόνο να σας μεταφέρω. Η Λουξεμβουργική Προεδρία θα έπρεπε να προσπαθήσει να επαναφέρει το πνεύμα της κοινοτική μεθόδου. Το περασμένο Σαββατοκύριακο συνέβη καταστροφή. Ό,τι προσπάθεια και να γίνει για να αποφευχθεί ο εκτροχιασμός, δύο στοιχεία της κοινοτική μεθόδου έχουν εξαφανιστεί πλήρως. Πρώτον, το ανώτερο συμφέρον που είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των εθνικών συμφερόντων και η προσπάθεια συμβίωσης των μεγάλων με τις μικρές χώρες και μεγάλες εννοώ και τη Γερμανία με την οποία θελήσαμε να κάνουμε συμφιλίωση. Ας μην επεκταθώ, θα ήθελα όμως και εσείς και ο Πρωθυπουργός σας τους επόμενους μήνες να κάνετε μια προσπάθεια στη δημόσια συζήτηση να πείτε μερικά πράγματα για να επαναφερθούν αυτές οι έννοιες που έχουν εξαφανιστεί. Ευχαριστούμε Σίλβια για την μεγαλειώδη σου παρέμβαση. Και τώρα ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Σμιτ για την παρουσία σας στην Επιτροπή μας, αλλά πάνω απ' όλα για, τους πολλούς, για τις πολλές που αναλάβατε εν ονόματι της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου. Συμφωνώ με τη Βιβιάν αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία που έχουμε αυτή την Προεδρία τώρα η οποία ιστορικά έχει δείξει πόσο πιστεύει στην ιστορική υπόθεση στην οποία και πολλοί από εμά πιστεύουμε. Το μόνο που θέλω να πω λοιπόν σε εσά είναι το θέμα της σημασίας που έχει μια απλή οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση. Πέρα από τις ελλείψεις των ενωσιακών πολιτικών, που είναι προφανείς, έτσι. Υπάρχει το θέμα, καταρχάς, της κοινωνικής διάστασης. Της δημοκρατικής διάστασης. Εκεί υπάρχουν ελλείψεις. Πέρα από τις ελλείψεις των πολιτικών, υπάρχει πάνω από όλα το πρόβλημα της διακυβέρνησης με την περιπλοκότητα που έχουν τα προβλήματα και με την οποία μπαίνουν τα προβλήματα, με την περιπλοκότητα της, ε, τη θεσμική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αδύνατον, είναι αβίωτο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τώρα και στο μέλλον. Όπως τέθηκε το θέμα της νομοθετικής απλούστευσης, η νομοθετική διαδικασία είπαμε ότι πρέπει να απλουστευτεί, με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο απλό έτσι και άμεσο τρόπο πρέπει να πούμε ότι πρέπει να πλουστευτεί και το θέμα της διακυβέρνησης. Το θέμα της νομοθετικής διαδικασίας το βλέπουμε με κάποια σύνεση και με φόβο. Οι διάφορε πολιτικέ ομάδε μεταξύ των οποίων και οι δικοί μου το βλέπουν έτσι με κάποιο φόβο, γιατί μπορούν, θεωρούν ότι μπορεί να είναι ένας μηχανισμός για να αποφύγουμε αποφάσεις κοινωνικού χαρακτήρα που θεωρούν ότι περιπλέκουν υποτίθεται την καλή λειτουργία της αγοράς. Και αυτή η λειτουργία της αγοράς πρέπει να λειτουργεί πιο απρόσκοπτα, δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιους, ε, τέτοιους, ε, τέτοιου τύπου παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, παρά μόνο καθαρά οικονομικού ας πούμε και ε, μερκαντιλιστικού. Εγώ θα έλεγα ότι πάνω απ' όλα πρέπει να απλουστευτεί ο θεσμικός μηχανισμός της Ένωσης. Και ακριβώς γι' αυτό σας ζητάω το Συμβούλιο, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, να μην είναι τόσο ανέστητο στις προτάσεις που εμφανίζονται για απλούστευση. Δεν θέλουμε να περιπλέξουμε την περαιτέρω τη διακυβέρνηση της Ένωσης. Παραδείγματος χάρη παράλληλο κοινοβούλιο των χωρών του ευρώ. Ένα συμβούλιο παράλληλο των χωρών του ευρώ. Και αν αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε για να πάρουμε μια απόφαση να, κάνουμε, να καταβάλουμε ανυπέρβλητες προσπάθειες, εάν περιπλέξουμε την πολιτική δομή της Ένωσης, πέραν το ότι θα έχουμε δημοκρατικές παρεμβολές, νομίζω ότι θα δίναμε και ένα χτύπημα την ε, πολιτική διακυβέρνηση τη Ένωση. Όπω είπε ένα γνωστό φιλόσοφο που όλοι ξέρουν, ο Μπέικον, είπε σε κάποια φάση ότι η αλήθεια μάλλον θα γεννηθεί από το λάθος παρά από τη σύγχυση. Και νομίζω ότι όλα αυτά που προκαλούν σύγχυση στο σύστημα πολιτικής διακυβέρνησης θίγουν τις πιθανότητες επιβίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μειώνουν τις πιθανότητες επιβίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άντερσον. Πρόεδρε, εκτιμώ ιδιαίτερα κύριε Υπουργέ το ότι ήρθατε στη δική μας την Επιτροπή. Αυτή εξ να σας πω κάτι που έχει σχέση με το πακέτο καλύτερη νομοθεσία. Εμείς οι πράσινοι ανησυχούμε. Ανησυχούμε για το ότι αυτό το θέμα, η καλύτερη νομοθεσία, στην πράξη, στην πρακτική σημαίνει χειρότερη νομοθεσία. Γι' αυτό το λόγο ελπίζουμε να μην υλοποιηθούν όλα αυτά. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι και σχετικά με αυτά που διαδραματίστηκαν το Σαββατοκύριακο. Από την σκοπιά της Σουηδίας, ε, την Οικονομική και Νομιζωτική Ένωση την ε, αντιμετωπίζουν οι Σουηδοί από κάποια απόσταση, αλλά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, αργά ή γρήγορα ενδέχεται κάποιες χώρες να επιλέξουν να βγουν από την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ανεξάρτητα τώρα αν το βρίσκει κανείς αυτό καλό ή κακό, κοιτάξτε, αν υπάρχει κάποια ε, συντεταγμένη έξοδος, αυτό ίσως είναι καλύτερο. Προφανώς και είναι καλύτερο, σίγουρα είναι καλύτερο από το να υπάρχει μια χαοτική έξοδος που κανείς δεν μπορεί να ξέρει τις συνέπειες. Εμείς λοιπόν ελπίζουμε η Προεδρία του Λουξεμβούργου να αρχίσει να τα σκέφτεται όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι που να θέλουν να υποβάλουν ερωτήματα... Θα ήθελα και εγώ να μου επιτρέψετε να κάνω μία ερώτηση στον Υπουργό. Κυρίως μία ερώτηση που αφορά στην κρίση που διερχόμεθα και που αφορά στην όλο και μεγαλύτερη έλλειψη κοινοτικής μεθόδου. Σήμερα αναφέρθηκε από τους Γκουλάρ, Καστάλλο, Σόλτς ότι είναι απαραίτητο να επανέλθουμε σε αυτή την κοινοτική μέθοδο. Και θέλω να εστιάσω την προσοχή μου σε ένα θέμα. Δεν πιστεύετε κι εσείς ότι είναι απαραίτητο να σκεφτούμε λιγάκι αυτή την εκπληκτικά ανώμαλη φύση που χαρακτηρίζει το Eurogroup. Εγώ παρακολούθησα όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα κατά τους ε, τελευταίους μήνες και διαπίστωσα ότι υπάρχει μια τεράστια δυναμία όχι μόνο στην κοινωτική μέθοδο αλλά και σε αυτό που λέμε rule of law, κράτος δικαίου. Ξέρετε γιατί, διότι συνέβη το εξής. Για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί ο Υπουργός ο Έλληνας αποκλείστηκε από συνεδριά του Eurogroup, προφανώς και αναφέρομαι στον Υπουργό κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος απευθύνθηκε στις νομικές υπηρεσίες ε, της ε, Ένωσης και η απάντηση του δόθηκε και παραθέτω είναι ότι εμείς ως Eurogroup δεν είμαστε νομικά κατοχυρωμένοι. Δεν υπάρχει καμία συνθήκη η οποία να έχει συστήσει το Eurogroup τέλος παράθεση. Άρα δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι βρισκόμαστε με ένα Eurogroup το οποίο δεν είναι υπόλογο σε κανένα. Ε, λειτουργεί μυστικά, ούτε καν πρακτικά δεν τηρεί των συνεδριάσεων που λαμβάνουν χώρα. Τώρα, για τους πολίτες, ξεχάστε τους πολίτες. πολίτες δεν ενημερώνονται σε τίποτα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι βρισκόμαστε όχι μόνο έξω από την κοινοτική διαδικασία, αλλά όλα αυτά δεν έχουν και καμία σχέση με αυτό που λέμε κράτος δικαίου και καμία σχέση με νομιμοποίηση λειτουργίας της Ευρωζώνης. Κύριε Υπουργέ, ε, τώρα πια έρχεται το λόγο για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ε, ερωτήσεις ή σε κάποιες από αυτές. Je Προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ε, απαντήσεις, μάλλον τις ερωτήσεις και θα απαντήσω ομαδικά σε κάποιες ερωτήσεις. Καταρχά για όλο το θέμα που αφορά την καλύτερη νομοθεσία, το better regulation. Καταλαβαίνετε δεν είμαι ο εκπρόσωπο του κ. Φερχόφστατ, πρώτα απ' όλα. Από ό,τι κατάλαβα θα τον προσκαλέσετε, θα τον ρωτήσετε, θα του δώσετε την εντολή που θέλετε να του δώσετε. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η πρώτη, στην πρώτη συνεδρία που κάναμε, την κάναμε για να οργανώσουμε τις εργασίες. Ήταν οργανωτικού χαρακτήρα. Ο κύριος Φερχόφστατ σας διαβεβαιώ ότι δεν ξεπέρασε τις ε, αρμοδιότητές του ή την εντολή του, εάν του δώσατε. Έχω, εν πάση περιπτώσει, εκπροσωπώ το Συμβούλιο και είναι δύσκολο να εκπροσωπεί κανεί το Συμβούλιο, πιστέψτε με. Δεν μπορούμε να ασχολούμε τώρα και με τα άλλα όργανα. Αυτό μας έλειπε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι, πρώτον, ότι όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε καλή νομοθεσία. Καλύτερη νομοθεσία δεν θέλει κανένα. Αδιαφανή νομοθεσία, υπερβολική νομοθεσία, εδώ αρχίζει να περιπλέκει το πράγμα. Δεν είναι όμορφο για την Ευρώπη όμως. Όταν περιπλέκονται τα πράγματα και όταν νομοθετούμε σε πράγματα που δεν πρέπει να νομοθετούμε, τα πράγματα χαλάνε. Συμφωνούμε εδώ, Προφανώ. Δεύτερον, και εδώ επίση είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται, δεν θέλουμε από το παραθυράκι να περιορίσουμε αρμοδιότητες που έχουν καθοριστεί από τις συνθήκες. Δεν θέλουμε τις νομοθετικές αρμοδιότητες που κατοχυρώνει η συνθήκη, δεν θέλουμε να τις περιστήλουμε. Αυτή η διαθεσμική συμφωνία, καθώς και όλα αφορούν την καλύτερη το έθνομοθετή, εν το better regulation, δεν πρέπει να ε, επηρεαστούν. Επίσης, οι πολιτικές πρέπει να έχουν την πρωτοκαθεδρία. Δεν είμαστε, ελπίζω, μία ένωση η οποία τις οποίες ηγείται, ε, ηγούνται τεχνοκράτες. Όχι, είμαστε πολιτική ένωση. Όχι ολοκληρωμένη κατά σέκατ εκατό άλλα πολιτικοί. Και οι αποφάσεις τελικά πρέπει να παίρνονται από του πολιτικούς. Δεν υπάρχουν λοιπόν φορεί, θεσμικά όργανα, χρήσιμες μερικές φορές, που ναι μεν σας δίνουν τη γνώμη τους, μπορεί να σας προειδοποιήσουν για τι συνέπειες κάποιων αποφάσεων, αλλά στην τελική, στο τέλο, στο κάτω-κάτω της γραφής, οι πολιτικοί παίρνουν τι αποφάσεις. Αυτή είναι η δημοκρατία. Έχουμε δύο κλάδους, Έχουμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στο νομοθετικό επίπεδο και αυτοί είναι οι δύο νομοθετικοί βραχίονες που παίρνουν τις αποφάσεις και τις ευθύνε τους. Η, η Κομισιόν πριν κάνει μία πρόταση, μια και έχει το μονοπόλιο έτσι, στην πραγματικότητα του δικαιώματος πρωτοβουλίας. Εκείνη αξιολογεί, ελέγχει, συνδιαλέγεται με τους ενδιαφερόμενους. Χρειάζεται κάτι τέτοιο. Αλλά τελικά πριτανεύει η πολιτική. Για ένα θέμα που με ενδιαφέρει τα μάλα, το κοινωνικό. Δεν μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να αποδομούμε όλα αυτά που έγιναν στο κοινωνικό επίπεδο. Πολλοί από εμά, και εγώ μεταξύ αυτών, θεωρούν ότι το κοινωνικό επίπεδο είναι ανεπαρκές στο οικονομικό πλαίσιο το σημερινό, της εσωτερικής αγοράς κτλ. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε τώρα μέσω του refit να ξεφορτωθούμε κάποια κοινωνικά στοιχεία. Έτσι. Και επειδή συζήτησα και με τον Επίτροπο Τίμερμαντς, πιστεύω ειλικρινά ότι δεν έχει την πρόθεση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σίγουρα όχι ο κύριος Τίμερμαντς. Λοιπόν, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Θα εργαστούμε ούτω ώστε να δούμε πώς μπορούμε οι, τα θεσμικά όργανα μπορούν να συνεργαστούν για τον πολιτικό, την πολιτική οργάνωση, για την αξιολόγηση των πολιτικών. Και εδώ επανέρχομαι σε κάτι που έκανε και το κοινοβουλίο πριν από 10 χρόνια. Τι είχαμε, ας πούμε, υπερβολικά πολλά νομοθετήματα. Από την υπερβολική νομοθεσία μπορούμε να περάσουμε στην υπερβολικά λίγη νομοθεσία. Πρέπει να δούμε και το κόστος αντίστροφα. Ποιο είναι το κόστος της μη νομοθεσίας, έτσι. Το κόστος της μη Ευρώπης, όπως έλεγε ο Ντελόρ, είναι το εξή ότι αν δεν έχουμε μια πραγματική Ευρώπη με κανόνες, όπου οι οικονομικοί φορείς ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ποια θα ήταν η συνέπεια. Θα ήταν προφανής θα, φτάσουμε, θα φτιάξουμε φραγμούς εδώ, φραγμούς εκεί, τροχοπέδι εδώ, τροχοπέδι εκεί και οι εταιρείε, ίσως όχι μεγάλες, αλλά οι μικρές, θα έχουν τρομερές δυσκολίες για να ανταγωνιστούν η μία την άλλη. Θα έχουν πάρα πολλά προβλήματα, θα, δεν θα μπορούν να πουλήσουν δεξιά και αριστερά, δεν θα μπορέσουν να παρέσχουν υπηρεσίε πέρα από τα σύνορά τους. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Και όλα αυτά, όλες οι συζητήσεις θα πρέπει να γίνουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα για τις μελέτες αντικτύπου. Ήμουν σαφής, χρειάζονται αυτές. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι πάνω από τις πολιτικές αποφάσεις. Πρέπει να το ξαναπούμε αυτό. Ακόμα μια φορά. Για τις εκλογέ. Με ρωτήσατε να σας εξηγήσω ότι είναι ο ρεαλισμός αυτό το πεδίο. Πάντα είναι δύσκολο να το εξηγούμε. Αλλά σίγουρα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές, κάποιες αλλαγές. Τους Εκλογικού νόμου. Εδώ είναι ένα θέμα εναρμόνιση. Είναι παράλληλο με αυτό, αντίστοιχο με αυτό που είπα προηγουμένω. Πρέπει να φτάσουμε σε λογικού, εναρμονισμένου κανόνε για το εκλογικό δίκαιο εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα. Όπου σε κάποιε χώρε για την άσκηση του βασικού δικαίωματος που είναι το δικαίωμα ψήφου τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. Για να πηγαίνουν από εδώ και πέρα πιο καλά. Όταν μιλήσαμε για, κάποιους, για είχαμε βρει ότι υπάρχουν πολύ μικρές, πολύ σφιχτές προθεσμίες σε κάποιες χώρες για να κατευθούν εκλογικοί κατάλογοι. Ένα μήνα, ας πούμε, σε κάποιες χώρες και σε κάποιες άλλες μία εβδομάδα. Γιατί, γιατί αυτές οι διαφορές. Θα πρέπει νομίζω εκεί να κάνουμε τις προσαρμογές αυτές και τις διορθώσεις κατάλληλες. Και είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με το κοινοβούλιο σας για να δούμε αυτά τα θέματα. Τώρα, για το μητρό αυτό τον λόμπι να το δούμε αυτό το θέμα. Είναι θέμα του Κοινοβουλίου σας όμως. Είναι και θέμα της Κομισιόν. Και εν μέρη είναι θέμα του Συμβουλίου. Αλλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για να συζητήσουμε τα πάντα και να εξασφαλίσουμε απόλυτη διαφάνεια ή όσο μεγαλύτερη διαφάνεια μπορούμε. Σε ό,τι αφορά την ΟΝΕ, και όλα όσα συνέβησαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Καταρχά, να μην σα δώσω την προσωπική μου άποψη, έτσι. Δεν έχω έρθει ε, ούτε ω Λουξεμβουργέζο Υπουργό, ούτε ω Νικολά Σμιτ. Είμαι εδώ ω εκπρόσωπο τη Προεδρία. Άρα θα πρέπει να σεβαστώ αυτό το ρόλο. Αυτό που είναι σαφέ και όλοι ξέρουν είναι ότι η οικοδόμηση της ΟΝΕ είναι απόλυτα ανεπαρκής. Έχουμε την έκθεση των πέντε Προέδρων και θα δώσω λιγάκι τη γνώμη μου εδώ. Σίγουρα πρέπει να βελτιωθούν κάποια πράγματα εκεί, έτσι. Κυρίως στο κοινωνικό επίπεδο. Και στο επίπεδο της θεσμικής λειτουργίας. Και αυτή είναι μια αρχή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες πολιτικές και άλλου τύπου, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή. Θα πρέπει να δουλέψουμε από αυτού. Σας είπα, αύριο μεταξύ των Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνει μία συζήτηση για την διακυβέρνηση και την τον τρόπο διακυβέρνησης του κοινωνικού, των κοινωνικών θεμάτων. Θα τα θέσουμε όλα αυτά επιτάπητος και θα σας ενημερώνω για τις συζητήσεις πάνω σε αυτή την έκθεση των πέντε προέδρων. Ο... Το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου της ΟΝΕ είναι ένα πρόβλημα, προφανώς. Δεν έχω λύση, δεν είναι και εύκολη. Ποιο θα είναι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα νέο σώμα. Ο συνάδελφος Α έφυγε είπε ότι δεν πρέπει να περιπλέξουμε περαιτέρω την λειτουργία των θεσμικών μας οργάνων. Συμφωνώ. Αλλά το πρόβλημα με το Eurogroup, και εδώ θα είμαι πολύ προσεκτικός, είναι απλό το πράγμα στην αρχή. Εγώ θυμάμαι τις παλιές συζητήσει. Δεν έπρεπε να υπάρχει πολιτική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Όλα ήταν στα χέρια της ΕΚΤ. Κακό είναι αυτό. Σήμερα βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μία νομισματική ένωση χωρίς πολιτική εξουσία. Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε μία πολιτική εξουσία πέρα από αυτό που ξέρουμε σήμερα ως ε, Eurogroup. Δεν πρέπει να υπάρχει το Eurogroup τώρα. Η πραγματικότητα, τα γεγονότα μας δείχνουν ότι κάποια προβλήματα της ζώνης ευρώ πρέπει να επιληθούν από τα, από τα μέλη της Ευρωζώνης. Τώρα έχουμε και ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρωζώνης. Εγώ θέλω να καλέσω τους υπουργούς εργασίας ε, της Ευρωζώνης για να συζητήσουν τα κοινωνικά θέματα της Ευρωζώνης. Γιατί όταν είμαστε σε μια νομισματική ένωση έχουμε διαφορετικού τύπου προβλήματα σε σχέση με αυτούς που δεν είναι στην ΟΝΕ, σε αυτή την Ένωση. Δεν θέλουμε να τους αποκλείσουμε, δεν είναι εκεί το θέμα. Πρέπει να τους ενημερώνουμε και να έχουμε στενούς δεσμούς. Αλλά όταν είμαστε σε μια ευρωζώνη, το είδαμε, έχουμε άλλα προβλήματα. Σε σχέση με αυτούς που δεν είναι στην ευρωζώνη. Για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων. σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ναι. Το Σεπτέμβριο θα είμαι έτοιμος να σας συναντήσω για να συζητήσετε θέματα που ενδιαφέρουν πολύ το Κοινοβούλιο. Ξέρετε όμως ότι παρότι με κολακεύει αυτό που λέτε για την Λουξεμβουργιάζικη Προεδρία, αλλά ξέρετε ότι η Προεδρία είναι απλώς η Προεδρία του Συμβουλίου. Δεν είναι ότι η Προεδρία του Συμβουλίου έχει την απόλυτη εξουσία στην Ένωση. Όταν κάτι με ρωτάει, όταν κάποιος με ρωτάει τι θα προτείνει η Προεδρία για την επικουρικότητα, δεν θα κάνει η Προεδρία προτάσεις. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε όσα υπάρχουν επιτάπητος και να βρούμε συμβιβασμούς. Γιατί ο ρόλος της Προεδρίας είναι να βοηθήσει τον κόσμο για να φτάσει σε συμβιβασμούς. Συμβιβασμούς στο Συμβούλιο, συμβου, ε, συμβασμούς ενδεχομένω και με τα άλλα θεσμικά όργανα και ενδεχομένως με το δικό σας. Βεβαίω μπορούμε να δούμε τις ανησυχίες που υπάρχουν, που Συμβουλίου λέει ο, ο αλλά μάλλον είναι του Κοινοβουλίου, σε ό,τι αφορά την Εκτεταστική Επιτροπή. Και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάποια σημεία ένωσης. Αλλά θα ήθελα να τα δούμε όλα αυτά ήρεμα, να δούμε πού έχουμε φτάσει, πού είμαστε και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το σημαντικό θέμα. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει να θεωρήσουμε αυτό το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής και αυτό το δικαίωμα που έχει το Κοινοβούλιο, το οποίο το έχει ως δικαίωμα. Δεν πρέπει να το θεωρήσουμε ως εχθρική πράξη απέναντι σε κάποιον, ποιον δηλαδή, την Κομισιόν, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη. Δεν θέλουμε να το δούμε έτσι. Το θέμα είναι αυτό το δικαίωμα που υπάρχει να το πλησιώσουμε από σαφείς κανόνες, ούτως ώστε να συμφωνήσει και το Συμβούλιο. Συμφωνώ επίσης με τα όσα είπε η Σιλβί Γκουλάχ, η οποία έφυγε. Το υπέρθετο συμφέρον. Μερικές φορές δυσκολευόμαστε να το βρούμε. Πού υπάρχει σε αυτές τις συζητήσεις γιατί είναι κάπου εκεί στις νεφέλες, γιατί τα θεσμικά όργανα κινούνται σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν, γιατί δεν είναι καλά οργανωμένα για να διαχειριστούν κρίσεις όπως αυτή που ζούμε. Είναι σαφές ότι όταν δημιουργήθηκε η ΩΝΕ, κανένας, και κακός βέβαια, κανένας δεν είχε φανταστεί. Ήμασταν σε, μια κατάσταση έτσι, μακαριότητας. Θεωρούσαμε ότι η κρίση όπως αυτή το 29 αποκλείεται να ξαναέρθει, να την ξαναζήσουμε. Και σήμερα ξέρουμε πολύ καλά ότι οι κρίσεις είναι πραγματικές και επανέρχονται. Και όπως αυτή που ζήσαμε μοιάζει με αυτή του 1929. Νομίζω τώρα ότι πρέπει να εργαστούμε για να ρυθμίσουμε, οργανώσουμε τα πράγματα. Και αυτό που υπόθηκε από τον Γιολάινεν για τα κράτη, τα μικρά και τα μεγάλα, για το εθνικό, την εθνική διάσταση που είναι πανταχού παρούσα, που δημιουργεί ασφυξία σε οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια έλλειψη σε επίπεδο εκπροσώπησης του υπέρτατου συμφέροντος, που είναι το ευρωπαϊκό συμφέρον. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να το προτάξουμε περαιτέρω αυτό το ευρωπαϊκό συμφέρον. που είναι τελικά μια κατάσταση νικηφόρα για όλους. Επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τα ΜΜΕ, ε, μερικές φορές αυτό το υπέρτατο συμφέρον λοιπόν χάνεται. Μια τελευταία λέξη. για την έξοδο από, το, από την Ευρωζώνη. Γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει η συνθήκη, οι συνθήκες. Ναι, βεβαίω θα πρέπει να αλλάξουν. Θα πρέπει να τα αλλάξουμε γρήγορα, δύσκολο. Ξέρουμε ότι οι χώρες οι οποίες θα κάνουν ε, δημοψηφίσματα είναι πολύ προσεκτικές. Αλλά υπάρχουν κενά στις ισχύουσες συνθήκες. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, προοδευτικά. Αν θέλουμε όμως η διαδικασία αυτή τελικά να στεφτεί από επιτυχία, χρειαζόμαστε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Γιατί αν δεν υπάρξει μια νέα εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, κάθε αναθεώρηση των συνθήκων θα αποτύχει στην Α ή στη Β χώρα. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί. Και δεν κερδίζεται με την αλλαγή των συνθήκων, αλλά με το τι σημαίνει η Ευρώπη για τους πολίτες, για τα κοινωνικά θέματα, για τα οικονομικά, για την προστασία του περιβάλλοντος κτλ. κτλ. Και ένα τελευταίο κοινοτική μέθοδος. Mm, ναι, βεβαίως. Είναι η μόνη που μας επιτρέπει να διαχειριστούμε το υπέρτατο συμφέρον, όπως είπε η Σιλβή. Είναι η μόνη που μας επιτρέπει να το εντοπίσουμε καλύτερα. Θα πρέπει να, το, να την αποκαταστήσουμε αυτή τη μέθοδο. Γι' αυτό θα πρέπει κάποια στοιχεία να τα επανεντάξουμε στο κοινοτικό πλαίσιο. Έτσι. Δεν μιλάω για τη συμμετοχή σε κάποιες διεθνείς, διεθνείς οργανισμούς, ε, κτλ. Δεν είναι και το θέμα. Αυτό που λείπει από την Ευρώπη είναι μια έντονη πολιτική διάσταση, το είπατε. Δεν μπορούμε να έχουμε μια νομισματική ένωση χωρίς να έχουμε μια πολιτική ένωση. Μα το είχαν πει στο παρελθόν. Πολλοί το είχαν πει. Ακόμη και αυτοί που ήταν κατά τη ΩΝΕ. Εγώ πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο του Φρίντμαν και όμως δεν είμαι θειασότης των οικονομικών θεωριών του Φρίντμαν. Είχε πει, εάν κάνετε μια νομισματική ένωση χωρίς πολιτική ένωση, θα διαλυθεί. Ορίστε. Και θα, θα δούμε και άλλες ρογμές, εάν δεν ενισχύσουμε την πολιτική ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για τις απαντήσεις σας. Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω ότι δεν υπήρχαν μόνο αισιόδοξοι μεταξύ των ιδρυτών του ευρώ. Υπενθυμίζω ότι ίσως γνωρίσατε τον κύριο Τομάζο Παντασκόπ που επεξεργάστηκε τα του ευρώ και είπε ρητά από την πρώτη μέρα του ευρώ ότι ένα νόμισμα χωρίς κράτος δεν μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα και σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα. Ευχαριστώ. Και καλό κουράγιο για την Προεδρία. Siamo arrivati al eh, penultimo punto, credo. No. Το τελευταίο σημείο νομίζω ή πρώτο τελευταίο. Είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και πιο συγκεκριμένα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους ε, στόχους εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί της πρότασης Ντάρικ Μακάλιστερ της γνωμοδότησης σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η γνωμοδότηση θα παρουσιαστεί όμως από τον κύριο Βίλαντ, γιατί η κυρία Μακάλιστερ δεν είναι παρούσα, δεν είναι εδώ και ζητάει συγγνώμη που δεν ήρθε. Είναι σαφές νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό γιατί ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών μετά ε, τον ψυχρό πόλεμο είναι πολύ σημαντικός. Σημαντικός ήταν κυρίως σε σχέση με τις στρατιωτικές παρεμβάσεις οι οποίες ε, έλαβαν χώρα και άσχετα από τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη είναι εκείνα που αποφασίζουν κατά πόσον θα εγκρίνονται πολιτικές παρέμβασεις ε, όπως αυτές ε, που αποφασίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σχέση με τη Λιβύη. Κύριε Βίλαντ, ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο να μας παρουσιάσετε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και να μας πείτε και τις δικές σας σκέψεις από αυτού του σχεδίου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Βίλαντ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ε, η συνάδελφος μακαλίστε, ο συνάδελφος με συγχωρείτε, μακαλίστε, με παρουσίασε να παρουσιάσω τη γνωμοδότηση αυτή γιατί είναι σε μια συνεδρίαση στην Ουάσιγκτον ε, και υπάρχει κάποιος ε, περιορισμός σχετικά με την έκθεση χρονικός. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος ε, Μακάλιστερ περιορίστηκε και στα πιο σημαντικά θέματα. Τα οποία θέματα αυτά είναι τα εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως ε, και με τη συνθήκη της Λισαμπόνας καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση στα Ηνωμένα Έθνη. Στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις που προτείνουν στα Ηνωμένα Έθνη, κυρίως στο ψήφισμα 65-276, όπου γίνεται λόγος για τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών στη λήψη αποφάσεων. Η συνεργασία και η συνοχή στα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να ε, ενισχυθούν περαιτέρω, έτσι ώστε να διατηρηθεί ειρήνη. Και αυτό που παίζει ρόλο είναι να ε, παρεμβαίνουν τα Ηνωμένα Έθνη διαμεσολαβητικά για να βελτιωθεί η όλη κατάσταση. Το τρίτο που είναι σημαντικό να λοιπόν υπάρχουν σταθερές σχέσεις ανάμεσα στα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι βασική προϋπόθεση για να διατηρηθούν οι τρεις πυλώνες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία και η ανάπτυξη. Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών ε, ενδείκνυται για να παρεμβαίνει στην, ε, στο παιχνίδι της ισορροπίας δυνάμεων. Ε, τα Ηνωμένα Έθνη οφείλουν να παρεύουν και στο θέμα της γραφειοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης, γι' αυτό λοιπόν επιθυμούμε να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος και διαφάνεια στα προγράμματα στήριξης. Εδώ είναι σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι πρέπει αυτό να ενημερώνεται για τις δαπάνες των Ηνωμένων Εθνών. Ο συνάδελφος Μακ Άλιστερ πέρα από αυτές τις ε, βασικές προϋποθέσεις έχει καταθέσει και διάφορες τροπολογίες ε, θεωρεί ότι πρέπει παραδείγματος χάρη να βελτιωθεί ή να βελτιωθεί το κομμάτι εκείνο που προβλέπει λεπτομέρειες για θέματα προϋπολογισμού, ελέγχου προϋπολογισμού και επίσης ε, θεωρεί ότι είναι σημαντικές κάποιες λεπτομέρειες που αποφασίστηκαν στις 2 Απριλίου του 2014 στην Ολομέλεια τότε υπήρχε μία σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται λοιπόν κυρίως για ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας, για να ενισχυθεί η νομοποίησή του, η περιφερειακή έκφρασή του, γιατί ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι να διεκδικήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έντρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Για να γίνει όμως αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω. Δηλαδή δεν είναι πια ε, τόσο εξελιγμένη η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να μιλούν με μία φωνή και μόνο αυτό αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο και η Γαλλία και η Αγγλία δεν θέλουν να παραιτηθούν από την έδρα του στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε λιγάκι το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ε, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο χάρτης ε, και να τεθεί το ερώτημα Ποιοι άλλοι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να αποκτήσουν επίσης ίδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρουσιάζεται ως αποτελεσματικός παίκτη, να μιλάει με μία μόνο φωνή και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν υπάρχει καλύτερη εναρμόνιση των θέσεων ε, των κρατών μελών και η ε, εναρμόνιση αυτών των θέσεων με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτά είναι τα βασικά σημεία τα οποία επισημαίνει ο συνάδελφος κύριος Μακάλιστερ και η διορία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 28 Αυγούστου. Αν έχετε ερωτήσεις, πολύ ευχαριστώ να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ. Γιολάιν. Mulțumesc, doamna președintă. Îi mulțumesc colegului meu, domnul McAllister, pentru un document foarte bun și cred că este un Ευχαριστώ τον κύριο Μακάλιστερ για το θαυμάσιο έγγραφο. Καλό σημείο θετηρία για τη συζήτηση. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. ω εισηγήτρια των σοσιαλιστών θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Καταρχά πρέπει να εξετάσουμε τη συνεργασία. Παλαιά μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΟΗΕ και μην ξεχνάμε και την χρηματοδότηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΟΗΕ που είναι σημαντική. Μην ξεχνάμε επίσης και ένα άλλο στοιχείο. Ο ΟΗΕ από το 1981 δεν είχε ε, ως Γενικό Γραμματέα κανέναν Ευρωπαίο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα να προτείνω ο επόμενο υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα να είναι ένας Ευρωπαίος. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε γυναίκα Γενική γραμματέα. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ. Θα ήθελα λοιπόν τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν μια, έναν Ευρωπαίο και μάλιστα Ευρωπαία ακόμα καλύτερα. Νομίζω ότι θα ήταν ένα σημάδι, ένα μήνυμα που θα στείλουμε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να προτείνουμε δηλαδή μια γυναίκα Ευρωπαία. Δεύτερον, όπως είπε και ο εισηγητής, η Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι ο πιο μεγάλος χρηματοδότης στο σύστημα του ΟΗΕ. Με βάση τα νούμερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τα 28 κράτη-μέλη πληρώνουν το 35% του προϋπολογισμού του ΟΗΕ και 36,8% ε, του προϋπολογισμού για την, τις εξωτερικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο του ΟΗΕ. Η, Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κράτη-μέλη μαζί δηλαδή ε, συνεισφέρουν ε, πάνω από 50% στα προγράμματα του ΟΗΕ που έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Είναι σημαντικό να συνεισφέρουμε στον προπολογισμό του ΟΗΕ και στα προγράμματα του ΟΗΕ. Αλλά έχω να κάνω παράλληλα μια παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλώς παρατηρήτρια. Δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Έχει πάρει ένα ειδικό καθεστώς, όντως. Δηλαδή, συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα σε πολλές διασκέψεις του ΟΗΕ. Όμως, αυτό το πράγμα δεν, δεν αντικατοπτρίζει το τη σημασία, το ειδικό βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την χρηματοδοτική της ε, συνεισφορά κτλ. Ως ε, εισηγήτρια, σκιώδη εισηγήτρια, θα το πω αυτό το θέμα για το κείμενο αυτό. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Το ψήφισμα 276 Θέλω να κάνει η Κομισιόν ε, μία μελέτη αντικτύπου για το ψήφισμα αυτό, για το κατά πόσο έχει εφαρμοστεί, τι διδάγματα έχουμε μάθει, για να έχουμε μία πολύ, καλή, πολύ καλύτερη πολυμερή προσέγγιση εκεί. Ευχαριστώ τον εισηγητή που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις μου και περιμένω τη συνεργασία για αυτό το θέμα. Πολύ ωραία. Ο κύριο Σόλτ, έχει το λόγο. <clears throat> Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την πρόταση που κατατέθηκε και θέλω να επισημάνω κάτι που είναι σημαντικό για μένα. Δηλαδή το ερώτημα, η δική μας Επιτροπή πού ακριβώς συμβάλλει νομίζω ότι στις εξηγήσει που ακούσαμε και στο αιτιολογικό ε, τη σκέψη, το αιτιολογικό το καταλάβαμε. Ε, αν σκεφτόμαστε με όρους εξωτερικής πολιτικής ε, ή αναπτυξιακής πολιτικής, αν σκεφτόμαστε τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη ή τη συμμετοχή καλύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική που χαράσουν τα Ηνωμένα Έθνη, εκεί συμφωνούμε. Υπάρχουν βέβαια πολλά θέματα που πρέπει να τα σκεφτούμε. Τι μπορεί παραδείγματος χάρη να βελτιωθεί στην πράξη. Όμως το ερώτημα που με απασχολεί εμένα είναι γιατί τελικά ασχολούμαστε εδώ στην Επιτροπή της Συνταγματικών Υποθέσεων με αυτό το θέμα. Ε, αφού το κάνουμε να πούμε το εξής και συμπληρώνω. Υπάρχει το ερώτημα του ποια είναι ακριβώς η εσωτερική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτή επηρεάζει τα ενωμένα Έθνη και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την επιρροή μας. Φτάνουμε λοιπόν στο ερώτημα που τέθηκε στην αρχή εναντί της ε, Προεδρίας. Είμαστε κάπου ανάμεσα σε μια οικονομική και νομισματική ένωση και σε μια μη εύρυθμα λειτουργούσα πολιτική ένωση. Αυτό είναι το έλλειμμα που υπάρχει γιατί αν θέλουμε να μας αναγνωρίζουν ως ένας αυτόνομος παίκτη, θα πρέπει και εμείς να πούμε ότι κοιτάξτε δεν είμαστε κράτος αλλά είμαστε ομοσπονδία κρατών. Οφείλουμε λοιπόν να το σκεφτούμε αυτό πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επηρεάζει κάποιες ε, πολιτικές ε, των ΗΕ, του ΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών και έτσι με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε μέσα στην ενίσχυση της επιρροής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, όσον αφορά τον είναι ε, Γενική Γραμματέας ε, των Ηνωμένων Εθνών Ευρώπη, σαφώς και τάσομαι ε, γυναίκα με συγχωρείτε, σαφώς και τάσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ αυτού. Πρόεδρος. Τι να, δεν λέω τίποτα για το τελευταίο, προφανώς. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Καστάλντο, στον Φάμπιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για να σκεφτούμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, αλλά τόσο περίπλοκο. Καταρχάς, γιατί και ως συντονιστή της Επιτροπής Εκτορικών Υποθέσεων είναι ένα μια στιγμή κρίση για την οργάνωση. Ο, ο ΙΕ είναι διαρεμένος. το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι διαιρεμένο γιατί ο κόσμος διαιρείται σε μπλοκ και αυτό είναι γεγονό. Όπως είναι γεγονό ότι και η δική μας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαιρεμένη σε μπλοκ. Και αυτό φάνηκε στις ελευθερές διαπραγματεύσεις για την ελληνική κρίση. Είναι παράδοξο που προσπαθούμε δηλαδή από τη μία, σωστά μεν, να έχουμε μια συνεπή θέση στο εσωτερικό του ΟΗΕ, αλλά το βασικό ερώτημα είναι μπορούμε εμείς να έχουμε αυτή την εσωτερική συνέπεια πριν προσπαθήσουμε να την υπερασπιστούμε στο εξωτερικό, στο εξωτερικό, στο εξωτερικό μας δηλαδή και απέναντι στον ΟΗΕ. Τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε δράσεις και συμπεριφορές που υποσκάπτουν και το ρόλο της ύπατης εκπροσώπου. Και δεν θα μιλήσω υποκριτικά, δεν κρύβομαι. Δεν θα, μείνω, δεν θα πω αοριστολογίες. Σα πω ένα παράδειγμα. Πρόκειται μια σοβαρή κρίση αυτή της Ουκρανίας. Και τελικά, Ποιο έπαιξε το ρόλο διαμεσολαβητή. Ποιο, Δύο αρχηγοί κρατών. Έτσι, ως συνήθως. Δύο από 28. Κάτι που εγώ θεωρώ όχι μόνο λάθος θεσμικός πώς. Γιατί υπάρχει και υπάρχει εκπρόσωπος έτσι, για ρόλο Και δεν θα έπρεπε καλώς να τη βοηθήσουν, να την ενισχύσουν, για να ενισχύσουν τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ειδικά έτσι πολύ χαρισματική ας πούμε αρχή κρατών και κυβερνήσεων. Αλλά να μην ξεχάσουμε ας πούμε την ε, κοινοτική θέση και τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι χάνει κύρος και έγκλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά τη όργανα, όταν πηγαίνει στι διεθνεί οργανώσει, α πούμε. Γιατί το ερώτημα που τίθεται έτσι και αυθόρμητα και στο εσωτερικό του ΟΗΕ είναι Α, και με ποιον πρέπει να μιλήσουμε για να δούμε ποια είναι η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ποιον, με την υπατή εκπρόσωπο, με κάποιο από τις πιο δυνα... κάποιον από τι πιο δυνατέ χώρε. Φυσικά είναι δράσει που έχουν επιπτώσει. Εμεί σίγουρα μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα τεχνικά βήματα στην Επιτροπή. Αλλά αμφιβάλλω πραγματικά ότι θα καταφέρουμε να έχουμε αποτελέσματα εξικέλευσα, εάν δεν εγγύθουμε πρώτα ότι η εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική και η κοινή ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, είναι η τελευταία λέξη. Έτσι. Έχουν αυτοί τον τελευταίο λόγο και είναι οι συνισταμένοι των εθνικών πολιτικών. Και μπορώ να σας δώσω ένα μακρύτατο κατάλογο περιπτώσεων όπου το εθνικό συμφέρον τελικά υπέσκαψε το υπέρτατο, πριτάνευσε. Μερικές φορές καταδικάστηκαν αυτά τα κράτη, άλλες φορές όχι. Τελικά αυτό ακυρώνει την κοινωτική μέθοδο, ακυρώνει το λόγο για τον οποίο δημιουργήσαμε αυτές τις πολιτικές. Νομίζω ότι κάποια δεν έγινε ακόμα πεταλούδα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει αυτή η συνέπεια. Ε, υπάρχουν και άλλοι επίσης, ε, άλλοι γεωπολιτικοί παράγοντες που μας επηρεάζουν στη δική μας, στο δικό μας γίγνεσθε και μας απομακρύνουν από το πραγματικά ευρωπαϊκό συμφέρον. Αυτά και θα παρουσιάσω σίγουρα τροπολογίες σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί αν δεν λύσουμε το πρόβλημα στη λύση του, δεν μπορούμε να λύσουμε και τα πρακτικά θέματα. Αν δεν λύσουμε το πρόβλημα στην, ε, στη ρίζα του, συγγνώμη, δεν μπορούμε να λύσουμε και τα βασικά θέματα. Και ελπίζω ότι κάποιο θα έχει το κουράγιο να πάρει μια θέση, να δώσει ένα μήνυμα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια, ούτω ώστε. Γιατί αν δεν έχουμε το κουράγιο να πούμε τα πράγματα ομά με το όνομά του, δεν θα βρούμε χρήσιμε λύσει και για την εικόνα μας, και για το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών που υπερασπιζόμαστε. Ευχαριστώ. Ε, grazie Fabio per le questioni che hai posto e per l'immagine anche del bruco e della farfalla. Credo che... Κοιτάξτε, πιστεύω ότι κάνουμε κατ' ουσίαν οπισθοχώρηση. Και κατ' ουσίαν επιστρέφουμε στις ε, εθνικιστικές ε, δυνάμεις της Ευρώπης που υπήρχαν και πριν από τον ε, ε, Παγκόσμιο Πόλεμο. L'onorevole Terry Cabras. Grazie, Presidente. Ε, ich werde wahrscheinlich ε, etwas ganz... Κοιτάξτε, εγώ θα πω ενδεχομένως... Ε, κάτι που μοιάζει με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Μακάλιστερ έθεσε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Και όσον αφορά το θέμα των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή, προέβαλε τις αδυναμίες που υπάρχουν σε επίπεδο θεσμών. Και ακριβώς αυτό διαρωτώ με. Πώς είναι δυνατόν να περιμένει κανείς ότι και με τον τρόπο αυτό από τις αδυναμίες δηλαδή θα προκύψει κάτι το αποτελεσματικό. Μα πώς πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να μην είμαστε αναγκασμένοι μετά από κάποια χρόνια να διαπιστώσουμε με απόλυτη θλίψη ότι τελικά δεν γίνεται τίποτα συζητάμε, συζητάμε, συζητάμε και δεν γίνεται τίποτα. Και άραγε τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε εν πάση τόσο κάτι να αρχίσει να κινείται σε αυτή την τόσο δύσκολη σχέση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εμείς ε, σας ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Αν δεν θέλει κανείς άλλος το λόγο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Βίλαντ. Όχι, κάποιος θέλει το λόγο ακόμα. Ο κύριος Λάινεν, με συγχωρείτε, δεν σας είχα δει, δεν σας είχα στον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Λάινεν. Το ερώτημα που ετέθη είναι τι ακριβώς ε, μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να συνεισφέρει αυτή εδώ η Συνταγματική Επιτροπή σε αυτήν την γνωμοδότηση. Νομίζω λοιπόν ότι στα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει σε σχέση με τα έθνη να τοποθετούμε τέτοια κριτήρια όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και δημοκρατικό έλεγχο. Θεωρώ ότι η έκθεση του κ. Μακάλιστα είναι καλή, αναφέρει κάποια χρήσιμα θέματα και πιστεύω πράγματι ότι η διαφάνεια των ΗΕ χρήζει βελτιώσεων. Ε, πολλά πήγαν στραβά και Όσον αφορά ας πούμε το θέμα του ελέγχου του προπλογισμού, εκεί πρέπει να γίνει μια σειρά από κινήσεις. Υπάρχει το θέμα της ε, αντιπροσωπευτικότητας. Αυτό το μόρφωμα πια είναι αναχρονιστικό. Δεν εκπροσωπεί και δεν αντιπροσωπεύει το κόσμο όσο έχει σήμερα. Και εν πάση περιπτώσει στο σημερινό κόσμο υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μια περιφερειακή ένωση. Μπορεί να προσθεθεί και η Ασιατική και η Αφρικανική Ένωση. Υπάρχουν και αυτές οι περιφερειακές ενώσεις. Έτσι λοιπόν αυτά τα ε, περιφερειακά σχήματα ε, θα πρέπει όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν ψήφο, δυνατότητα να είναι πλήρη μέλη και όχι μόνο παρατηρητές. Παραδείγματο χάρη ε, στην συνθήκη για το κλίμα, εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και έδρα και ψήφο. Δεν είναι απλώς παρατηρητής. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι στο Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να εμφανίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε πολύ καλά βέβαια ότι υπάρχουν δύο ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κέντρα και ψήφο. Αν όμως τελικά διευρυνθεί αυτό το σχήμα των Ηνωμένων Εθνών πρέπει η Ευρωπαϊκή ναι. Ένωση να αποκτήσει τέτοια δικαιώματα γιατί υπάρχει συνθήκη της Λισαβόνας που λέει ότι όλα τα κράτη έχουν κοινή εξωτερική πολιτική. Αυτός είναι τουλάχιστον ο στόχος. Όσον αφορά τώρα το δημοκρατικό έλεγχο, πολύ εξημών είμαστε υπέρ ε, της εκστρατείας που λέει ε, υπάρχει κοινοβουλευτική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι ο εισηγητής στο σημείο υπαριθμών 1 μιλάει για ένα παγκόσμιο κοινοβούλιο, το οποίο βέβαια είναι μια πολύ πομπόδης λέξη και αν θέλετε η δική μας η εκστρατεία ε, μιλάει για κοινοβουλευτική συνέλευση που θα ξεκινάει όπως ακριβώς ξεκίνησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή ένα είδος συμβουλευτικού οργάνου το οποίο θα απαρτίζεται από αντιπροσωπείες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, λοιπόν, επί της ουσίας, το άρθρο 1 της έκθεσης κατά άποψή μα είναι εντάξει, αλλά εγώ θα καταθέσω μία τροπολογία που θα αφορά στο δημοκρατικό έλεγχο των κοινοβουλίων των κοινοβουλίων των κρατών μελών των εθνών, Προφανώς αυτά είναι τα εθνικά κοινοβούλια και αν αποκτήσουμε και εμείς έντρα και ψήφο θα αφορά έλεγχο και σε εμά. Εγώ το βρίσκω πολύ αναχρονιστικό το να λένε τα Ηνωμένα Έθνη. Ξέρετε και οι ΜΚΟ έχουν ε, κάποιο καθεστώς αλλά όχι οι εκπρόσωποι των πολιτών. Ε, η Greenpeace, η Amnesty International, αυτοί όλοι είναι απλοί παρατηρητές. Τι είναι αυτό. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί, αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον. Ευχαριστώ. Γιώ. Φλιβερό το ότι πρέπει να συζητάμε ακόμα τη δυνατότητα εκπροσώπησης στο Συμβούλιο ασφαλεία. Ενώ θα έπρεπε εδώ και χρόνια να το έχουμε εξασφαλίσει. Κύριε Βίλαντ, μπορείτε να καταλήξετε σε κάποια συμπεράσματα. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να μεταφέρω και θα το μεταφέρω στον εισηγητή ότι είναι ένας... Ε, υπήρξε και ένας διερμηνέας, ε, με ένας βουλευτής που δεν είναι Γερμανός και μίλησε μάλιστα ε, τοπική διάλεκτο της Γερμανίας. Τέλος πάντων. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν ήταν... Ε, πολύ σημαντικά και όλοι προβληματίστηκαν για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο να ζητάμε μία έδρα και μία φωνή και, μία, και ψήφο τη στιγμή που μόνοι μας δεν έχουμε συμφωνήσει πώς θα το κάνουμε αυτό. Ίσως πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τους δικούς μας τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων πριν τελικά αποκτήσουμε κάτι που δεν θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει, δεν ε, οικειοποιούμε το ρόλο του εισηγητή, αλλά αυτό που είπε ο κ. Σόλτς, παρόλα αυτά, θέλω να το χαρακτηρίσω ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Δηλαδή, να δούμε λιγάκι ε, ποια είναι τα προγράμματα, τα projects ε, που τρέχουν στα Ενωμένα και ίσως να επιμείνουμε με τα δικά μας τα χρήματα να υποστηρίζουμε τα προγράμματα εκείνα τα οποία θεωρούμε αποτελεσματικά γιατί με τον τρόπο αυτό δεν είναι μόνο θέμα διαφάνειας να βλέπουμε δηλαδή τι γίνεται με τα δικά μας τα χρήματα αλλά με αυτόν τον τρόπο θα καλέσουμε και άλλους να πετήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Τώρα είναι λιγάκι αυτή η πρώτη μου αντίδραση αυτό που ελέγχθη σχετικά με την κοινοβουλευτική διάσταση και την κοινοβουλευτική συνέλευση. Έτσι, πρώτη απάντηση που μπορώ να δώσω είναι, είναι λίγο δύσκολο κοινοβουλευτική συνέλευση των δικτατόρων. Γιατί υπάρχουν και τέτοια κράτη που έχουν τέτοιο καθεστώς και πώς θα συμμετέχουν αυτά. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Καστάλτο. Θα το κουβεντιάσω αυτό ε, με τον εισηγητή, τον κύριο Μακάλισε. Κοιτάξτε, το παρελθόν μπήξε κάτι που πήγε πολύ καλά. Δηλαδή, αυτή η κοινοβουλευτική διάσταση στο θέμα της ε, πληροφορικής, εκεί ε, κάπως τα κατάφερε να καταξιωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, Εκεί έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η Ιταλία. Βέβαια το πρόγραμμα κάπου κόλλησε και νομίζω ότι όσον αφορά την ψηφιοποίηση και την πρόσβαση του πολίτη στο κοινοβούλιο του μέσα από το διαδίκτυο, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project που πρέπει να το στηρίξουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι όπου υπάρχουν ε, μέσα κοινωνική δικτύωση ότι και έχουμε και καλύτερη δημοκρατία. Κάθε άλλο, δεν το λέω αυτό. Αλλά λέω ότι η συμμετοχή του πολίτη μέσα από αυτά τα δίκτυα όπου υπάρχει δημοκρατία οδηγεί σε μεγαλύτερη σταθεροποίηση. Αυτό λέω και ίσως πρέπει λιγάκι να το δούμε αυτό το θέμα. Τώρα, να υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα για το σημείο. Να σας πω τρεις ημερομηνίες. 28 Αυγούστου 28 Αυγούστου του 15 μέχρι τις 12 η ώρα λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες. Όχι. Όχι, όχι. Ναι. 28 Αυγούστου, 12 ε, το μεσημέρι, πέφτει η Λεμιτόμος. Για να μπορέσετε να ψηφίσετε μετά στις 22 Σεπτεμβρίου, φέτος, το 2015, για να εξετάσουμε λοιπόν τις τροπολογίες και να τις ψηφίσουμε. Συμφωνείτε. Και πάμε στο τελευταίο σημείο. Πρόταση κανονισμού. Επιστρέφουμε στο σημείο ε, το οποίο είχαμε θίξει ήδη για την πρόταση κανονισμού για τους τρόπους και τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αντικαθιστά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 19 η Απριλίου του 1995. Ο εισηγητής είναι ο Ραμόν Χαουρέγγι Ατόντο. Δεν θα μακρηγορήσω εξηγώντα το θέμα. Γιατί ούτως ή άλλως έχουμε αρχίσει να συζητάμε. Ε, και το συζητήσαμε με την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Τώρα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι η τελευταία σας παρέμβαση στην ΑΦΚΟ ήταν στις 5 ε, Μαΐου. Και μπορώ να φανταστώ ότι θα μας ενημερώσετε κυρίως για δύο θέματα, κύριε Χαουρέγγι, δηλαδή ε, η συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 5 στην τελευταία πέμπτη, την πέμπτη που μας πέρασε και θα μας ενημερώσετε και για το τι ακριβώς προέκυψε ε, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Γενικών Υποθέσεων του Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω το λόγο για να μερώσετε για τα θέματα αυτά. Σύντομα. Θα ήθελα πρώτος, πρόεδρος Χιούμπνερ να βάλει στην ε, ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας τη δυνατότητα να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής ΑΦΚΟ για την κατάσταση, για το πώς έχουν τα πράγματα. Γιατί τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου δημιουργήθηκε ένα διέξοδο και θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής για τις εξελίξεις του θέματος αυτού. Να σας υπενθυμίσω πώς έχει το θέμα, πώς έχουν τα πράγματα. Εν μέρη το ανέπτυξα όταν απευθύνθηκα στο, στη στην Προεδρία. Έχουμε ε, μία έκθεση που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το 2013 του David Martin που ολοκλήρωνε, που ήταν το τελευταίο σημείο μιας διαπραγμάτευσης που δεν κατέληξε με συμφωνία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν γιατί δεν υπήρξε συμφωνία με αυτά τα δύο όργανα. Το Κοινοβούλιο το ενέκρινε για να μην καταπέσει και στην αρχή αυτή της νέας κοινοβουλευτική θητεία κληρονομήσαμε, εν την έκθεση αυτήν την κατάσταση. Η Επιτροπή ΑΦΚΟ και η πρόεδρος Χιούμπνερ ζήτησε από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν να ξεκινήσει ένα διάλογο για να έτσι, έχουμε μια νέα επαφή μαζί τους και τι είναι σίγουρο τώρα, σε όλη αυτή την περίοδο που έχει εκπνεύσει από το πρώτο, δηλαδή όλο αυτό το πρώτο εξάμεινο, εν πάση τη Ηλεκτρονική Προεδρία, με την οποία συζήτησα πολλέ φορέ, ανταλλάξαμε και επιστολέ. Πού καταλήξαμε, Καταλήξαμε να, κάνουμε μία συνεδρίαση 18 Ιουνίου με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο. Ε, θα ήταν άτυπη συνεδρίαση, τεχνική και διερευνητική γιατί το Συμβούλιο δεν είχε εντολή για να διοργανωθεί μια συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Ώρες πριν από τη συνεδρίαση αυτή που είχαμε συγκαλέσει εδώ στο Κοινοβούλιο, με τους εισηγητές, με τις ομάδες της κλασικές, με τις ε, νομικές υπηρεσίες της κάθε πολιτικής ομάδας, ώρες πριν, η Λετωνική Προεδρία μου έστειλε ένα email και μου επιβεβαίωσε ότι δεν μπορούσαν να έρθουν στη συνεδρίαση αυτή, το Συμβούλιο. Γιατί, γιατί το Συμβούλιο... Στο Συμβούλιο υπήρχε μία ε, μειοψηφία ανασχετική κατά τη συνεδρίαση αυτή. Στο μεταξύ υπήρχε μια νέα νομική γνωμοδότηση του Συμβουλίου για τις ε, τεχνικές αντιρρήσεις και πολιτικές αντιρρήσεις που έχει το Συμβούλιο απέναντι στην έκθεση David Martin και που έπρεπε να μελετήσει υποτίθεται το Συμβούλιο πριν από την συνεδρίαση αυτή που θα κάνουμε. Εγώ θα ζητούσα, εγώ ζήτησα μάλλον ε, στην εκπρόσωπο τη Λεπτονική Προεδρία να έρθει την επόμενη ε, μέρα για να το εξηγήσει. Γιατί όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών νομών θα ήταν εκεί και θα ερχόταν και η Κομισιόν ούτω ή άλλω στην συνεδρίαση αυτή. Και έτσι συνέβη. Ε, συνεδρίασα με την Λουτωνική Προεδρία στις 18 Ιουνίου ήρθε ως παρατηρήτρια και είδε την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου για τα προβλήματα που είχαμε σε αυτή την έκθεση. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε αυτή την έκθεση είναι ευέλικτος. Πάντα προσπαθούμε να βρούμε συμφωνία και με βάση τις διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει πριν από την έγκριση του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, πριν να έγιναν ε, διαπραγματεύσει επί 1,5 χρόνο στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, που δεν κατέληξαν σε 100% συμφωνία, αλλά ε, υπήρχε συμφωνία για πολλά από τα άρθρα τη έκθεση. Τώρα, τι συνέβη από εκεί πέρα. Η διαμαρτυρία μας και ο τρόπος με τον οποίο το Συμβούλιο βλέπει ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα και θέλουμε να συζητήσουμε, ανάγκασε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να αναλύσει. Μέχρι ποιο, ποιου σημείου το Συμβούλιο θα μπορούσε να μείνει στο περιθώριο. Ένα τέτοιο διαλόγο που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Και με θλίβει που το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή ετοιμάζει μια επίσημη απάντηση στην ε, πρόεδρο της ΑΦΚΟ, τη Χιούμπνερ, για να της μιλήσει για την ε, θέλησή του για το διάλογο αυτό. Υποτίθεται, με βάση τα όσα έμαθα και που τα επιβεβαίωσε ο ο Υπουργό, μα είπε, έμαθα ότι ο, το Συμβούλιο δεν θα θέσει άλλα εμπόδια στο διάλογο. Ε, αλλά μου είπαν ότι έχουν πάρα πολλέ νομικέ και πολιτικέ αντιρρήσει. και που θέλουν να εκφράσουν ε, και που θα τι εκφράσουν με, μια νέα έκθεση. Μα λείβει αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά νομικά και πολιτικά προβλήματα και αντιρρήσεις για την ε, έκθεση που είχε εγκρίνει το Κοινοβούλιο του Μάρτιν. Αλλά το καλό νέο που μας το επιβεβαίωσε ο υπουργό είναι ότι τελικά η Προεδρία του Λουξεμβούργου θα δεχθεί αυτό το διάλογο τουλάχιστον αρχικά. ότι θα κάνουμε αυτή την τεχνική διερευνητική mm. συνεδρία και να δούμε πού υπάρχει το πρόβλημα. Αν τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει θέληση διαπραγματεύση. τότε ναι, τότε θα πρέπει να πάρουν εντολή διαπραγμάτευση. Και εμεί, βεβαίω, το Συμβούλιο θα πρέπει να πάρει τέτοια εντολή, και εμεί θα δούμε τι μέθοδο εργασία θα έχουμε ε, σε αυτό το διάλογο με την Κομισιόν ή στον τριμερή διάλογο με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Αυτά. Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να ενημερώσω τα διάφορα μέλη τη Επιτροπή για το πώ έχουν τα πράγματα. Θεωρούσα ότι είχαμε φτάσει σε αδιέξοδο, αλλά ευτυχώ τελικά βλέπω ότι ο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα εγκρίνει μια επιστολή αποδοχή του διαλόγου και ο Λουξεμβούργιος υπουργό με τον τρόπο του το επιβεβαίωσε και το Σεπτέμβριο θα ξαναρχίσει αυτός ο διάλογος και θα σας ενημερώσω για τις όποιες εξελίξεις. Ευχαριστώ. Μα, και... Ε, θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ ε, εντυπωσιάστηκα από τις ε, αντιδράσεις ε, της νέας Προεδρίας, εντυπωσιάστηκα θετικά μετά από αυτό τον αποκλεισμό που είχε ασκηθεί από την προηγούμενη Προεδρία. Άρα δηλαδή το βρήκα, βρήκα αυτή την αντίδραση του Συμβουλίου ενθαρρυντική. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, κύριε Ατόντο, και την πρόεδρο η οποία επιμένει σε αυτό το θέμα γιατί σε τελική ανάλυση αν ε, επιμείνει θα και... Στο σημείο αυτό κατ' ουσίαν τελειώσαμε μισό λεπτό, μισό λεπτό τελειώσαμε ακόμα γιατί πρέπει να αναφέρω ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο πρέπει να εγκρίνεται και μισό λεπτό. Α, δεν χρειάζεται. Καλά. Δεν χρειάζεται, το έχετε πάρει ήδη το χρονοδιάγραμμα. Μου είπαν ότι δεν χρειάζεται. Εγώ νόμιζα ότι χρειάζεται, τέλο πάντων. Ε, τώρα σας εύχομαι καλές διακοπές, να περάσετε καλά. Και η επόμενη συνεδρίαση Θέλετε να ξέρετε πότε θα είναι η επόμενη. Θα είναι την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 3 ε, το απόγευμα μέχρι τις 6.30 εντός Φερξέλλης. Γεια Ο τραλε 15 18.30. E e Από 3 με, 6.30. Successiva volete fare silenzio Για την επόμενη, παρακαλώ, μπορείτε να σχάσετε, μπορείτε να ρεμίσετε λιγάκι. Seconda riunione lunedì. Δεύτερη, Δευτέρα. 21, α, τα ξέρετε αυτά. 21 Σεπτέμβρη. 21 Σεπτεμβρίου 2015. Buone vacanze. Grazie, grazie, grazie. grazie. Ha rianimato questa commissione, ha rianimato questa commissione.